Mes chers collègues, je vais vous demander... Αγαπητοί συναδελφοί, θα ήθελα να καθίσετε. Καλημέρα σας. Υπάρχει κάμερα γιατί θα γίνει αναμετάδοση από την Ολλανδική τηλεόραση και χαιρόμαστε να σας καλωσορίσουμε στην συνεδρίασή μας. Λοιπόν, αρχίζουμε. Ανακοινώσεις της Προέδρου για τις αποφάσεις των συντονιστών. Θα βρείτε τα αντίτυπα, το αντίτυπο τη συνεδρία της 25 Σεπτεμβρίου και της 11 ε, Οκτωβρίου. Έχουν διανεμηθεί τα έγγραφα. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέχρι το 12.30 θα θεωρήσουμε ότι οι αποφάσεις γίνονται αποδεκτές. Τώρα περνάμε στις ψηφοφορίες. Πριν όμως από την έναρξη θα Ήθελα να ξέρω αν ε, έχουμε απαρτία. Λοιπόν, επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ωραία. Όλα βαίνουν καλώς. Αρχίζουμε λοιπόν με την έκθεση ΚΟΧ, Διάσωση Ζωών, Ενίσχυση Ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκθεση πρωτοβουλίας. Αρχίζουμε λοιπόν. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αποδεκτή. Διακόπτη πρόεδρος. Τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Άρχεται η ψηφοφορία. Επαλήθευση. πέρας. Η τροπολογία απορρίπτεται. Τροπολογία 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές ε, αποδεκτή 35. Τροπολογία 36. Θέλετε παλήθευση, εντάξει. Άρχεται η ψηφοφορία για την 35. Πέρας. Εγκρίνεται η 35. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 38 υπέρ. Αν θέλετε παλήθευση και για την 36. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία για την 36. Πέρας. Ισοψηφία. Άρα απορρίπτεται. Δυστυχώς απορρίπτεται. Τροπολογία 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 Τροπολογία 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Επαληθεύουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται η ΕΠΤΑ. Τροπολογία 70, υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την 70, πέρας, η 70 εγκρίνεται. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ήμκο 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Ήμκο 18. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήμκο 18. 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 74 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 75 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, η 76 εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές ή 80 εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές επαληθεύουμε ηλεκτρονικά για την 84 πέρας. Απορρίπτεται η 84. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 97 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. 98-99 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 100. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Κύριε Βίμ Βαντεκάμπ, ε, καταψηφίζετε τις δικές σας τροπολογίες. Ο καθένας κάνει βέβαια ό,τι θέλει. Δικό σας θέμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές ή 101 απορρίπτεται. 102 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 103. Α, όχι, όχι, όχι. Δεν την ψηφίζουμε. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 106. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές η συμβιβαστική 11 εγκρίνεται. Ήμκο 16. Όχι, καταπίπτει. 119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 κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 147 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 148 υπέρ. Κύριε Βαντεκάμπ, δεν αγαπάτε τις τροπολογίες σας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 148. Θέλετε παλήθευση, ωραία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Κύριε Ερτούγκ, έχετε δίκιο. Η 148 εγκρίνεται, παρόλο που ο κύριος Κάμπ καταψήφισε. Ευτυχώς που είστε εδώ, κύριε Ερτούγκ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συμβαστική 18 υπέρ. Καταπίπτει η 149 διότι εγκρίθηκε η 148. Κύριε Ρικέ, καταλάβατε θαύμα. Συμβαστική 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 178 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 179 υπέρ. Κατά Αποχές η 179 εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 197 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 200 υπέρ κατά αποχές η 200 εγκρίνεται 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 202 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 204 υπέρ δεν θα κάνω πλέον σχόλια για τον κύριο Βαντεκάμπ. 204 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 205 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θέλετε επαλήθευση, ωραία, επαληθεύουμε, άρχεται η ψηφοφορία πέρας. Απορρίπτεται η 205. Συμβαστική 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 214. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 216. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 217 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 219 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία α θέλετε έλεγχο ωραία ελέγχουμε την 20 πέρας εγκρίνεται τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το σχέδιο έκθεσης, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. 43 υπέρ, ένας κατά και μία αποχή. Μπράβο σας, κύριε Κόχ. Ευχαριστώ του συνάδελφου. Allez, nous Περνάμε τώρα στην έκθεση Λούγκρεν σε σχέση με τους οδηγούς ορισμένων οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών και άδειες οδήγησης. Ωραία, αρχίζουμε. Δύο, Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ένα, Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έχουμε δύο ταυτόσημες, 48-49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε δύο ταυτόσημες. Α, όχι, όχι, καταπίπτουν. Με συγχωρείτε γιατί εγκρίναμε την 11. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με την 63 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Θέλετε Επαλήθευση κύριε Ερτούγκ. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία για την 63. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Έχετε δίκιο. Εγκρίνεται. Σαράντα. Υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά θα επαληθεύσουμε καλύτερα αρχίζει η ψηφοφορία για την 40 πέρας πράγματι εγκρίνεται εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 73. Α, όχι. Ως προς τη σύνταξη δεν, δεν, δεν την ψηφίζουμε. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ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 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26, έξι υπέρ όχι όχι όχι λέει η γραμματεία Ψηφίζουμε την 26 πέρα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27. Καταπίπτει γιατί υπερψηφίσαμε την 26. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά, αποχές, δεν είναι σαφές. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται με πλειοψηφία μεγάλη. 33 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε παλήθευση, εντάξει. Άρχεται η ψηφοφορία για την 35. Πέρας. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38. Υπέρ. Κατά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 κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το τελικό κείμενο ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 47 καμία ε, αποχή και καμία ψήφος κατά. Μπράβο, κύριε. Μπράβο σας κύριε Λούγκριν. Ομοφωνία. Συνεχίζουμε. Υπέρ ή κατά των διαπραγματεύσεων. Θα μας δώσετε εντολή ηλεκτρονικά υπέρ. Κατά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Πέρας, πέρας τώρα. 44 υπέρ και κατά δύο. Έχετε λοιπόν την εντολή ε, διαπραγματεύσεων. Μπράβο σας κύριε Λούγκρεν. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με την έκθεση Λούση Άντερσον για τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων. Έχουν αποσυρθεί οι δύο πρώτες τροπολογίες. Αρχίζουμε με την 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 205. Θέλετε επαλήθευση. Ωραία. Ηλεκτρονική για την 40. πέρας. Έχετε δίκιο, εγκρίθηκε. 205. Α, όχι, όχι, καταπίπτει. Συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία για τη συμβιβαστική 23. Υπάρχει αντίρρηση ως προς αυτή την προφορική. Υπάρχει αντίρρηση, φαίνεται πως όχι, άρα ψηφίζουμε. Υπέρ. Συμβιβαστική 23 στο σύνολό της υπέρ. 23, ναι, ναι υπέρ, υπέρ, της 23, της συμβαστικής, κατά. 23 ψηφίζουμε. Συμβαστική 23. Βαντεκάμ. Καρίμα. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ξεχωριστά την προφορική. Ωραία, θα ψηφίσουμε τη συμβαστική 23 που συμπεριλαμβάνει την προφορική. Δεν υπήρξαν αντιρρήσεις για την προφορική. Άρα εντάσσεται στη συμβιβαστική. Ψηφίζουμε την 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, προχωράμε αρκετά γρήγορα. Συμβαστική 6 υπέρ. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άρα θα δούμε κάθε τροπολογία χωριστά. Σε πρώτη φάση έχουμε τις τροπολογίες 66 έως και την ΙΜΚΟ 66 είναι υπέρ του συνόλου αυτών των τροπολογιών κατά εγκρίνονται. Και περνάμε στην συμβιβαστική εννέα Συμβαστική εννέα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 90 υπέρ. Κατά αποχές η 90 εγκρίνεται. Συμβαστική δεκα, ε, ε μάλλον 88 υπέρ. Κατά αποχές η 88 απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε επαλήθευση. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται με 29 υπέρ. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 89. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 158 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 158 συμβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 5. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Άρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά 109. Πέρας. Είναι σαφές ότι δεν ήταν σαφές, λέει η Πρόεδρος. Άρα απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά της συμβαστικής αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε επαλήθευση. Ωραία, επαληθεύουμε την 119. Πέρας. Εγκρίνεται η 119. Συμβαστική 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 13. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 133 συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήμκο 20. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΙΜΚΟ 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 25 υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά θα ήθελα να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας Απορρίπτεται, πράγματι. Ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά για την τελική έκθεση όπως έχει τροποποιηθεί, πέρας. ...43 ψήφοι υπέρ, 3 κατά. Κυρία Λούση Άντερσον, εγκρίνεται η εκθέσή σας. Και τώρα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την εντολή διαπραγμάτευσης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 42 υπέρ. Ναι, έχετε εντολή διαπραγμάτευσης. Συγχαρητήρια κυρία Άντερσον. Πάει και αυτό. Θέλετε το λόγο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ συνάδελφοι και θα ήθελα να σας πω ότι θα λάβω αυτή την εντολή και θα τα λάβω όλα αυτά υπόψη μου. Ε, ναι, σίγουρα αυτό θα προσθεθεί ε, στην ημερήσια διάταξη της επόμενης Ολομέλειας. Ωραία, το καταγράφουμε. Και συνεχίζουμε με την επόμενη έκθεση που είναι η έκθεση του κυρίου Eichhout Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Κινητικότητα Χαμηλών Εκπομπών. Είσαστε έτοιμοι. Έχουμε 59 σελίδες. Ωραία, ξεκινάμε. Συμβαστική 1, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ωραία, θα επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 73. Πέρας. Απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Θέλετε να επαληθεύσουμε. Ωραία, επαληθεύουμε. Ψηφίσατε όλοι. Για την 75. Πέρας. Εγκρίνεται, γι' αυτό είπα νομίζω. MV47 υπέρ κατά η MV47 εγκρίνεται 89 υπέρ κατά αποχές εδώ είμαι σίγουρη ότι απορρίπτεται 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. MV38. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έχουμε μια προσθήκη στη συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεν εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 8. Ωραία, άρχεται η ψηφοφορία αφού θέλετε να επαληθεύσουμε για την συμβαστική 8. Πέρας. Εγκρίνεται συμβαστική 8. 120. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εκατόν τριάντα Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ωραία. Επαληθεύουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 136. Εγώ νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Πέρας και πράγματι απορρίπτεται. 137 υπέρ. Α, διστάζεται κύριε Βαντεκάμπ κατά. Αποχές η 137 απορρίπτεται. 138 υπέρ. Τα αποχές εγκρίνεται. Νομίζω ότι ήταν σαφές, εν πάση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ήταν σαφές. Υπέρ 23, άρα εγκρίνεται. Συμβαστική 9, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εκατόν υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές, ξαναρχίζουμε. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές Τώρα είναι σαφές, συγκρίνεται. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 184 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται. Εκατόν έξι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 186 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Θέλετε επαλήθευση, ωραία. Ψηφίζουμε για την 190 ηλεκτρονικά. Πέρας. Είχε... Είχατε δίκιο. Είχατε δίκιο. Με μικρή διαφορά εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 196 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 197 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έμβη 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. πίσουμε τον υπότιτλο παραγράφου υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. MV8 υπέρ. Α, δεν είναι καθόλου σαφές. Υπέρ. MV8 υπέρ. Κατά. Θα υπαλληθεύσουμε γιατί πολύ δεν σηκώνετε το χέρι σας. Άρχεται λοιπόν πέρας για την MV8. Τώρα είναι σαφές το αποτέλεσμα. Συμβαστική 15α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 15α εγκρίνεται. 15 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 211 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 229 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 230 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 231 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 233 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Λοιπόν, καταπίπτουν τα υπόλοιπα και περνάμε στην έμβη 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θα επαληθεύσουμε έμβη 48 Allez, je ferme le vote. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Έμβη 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 243. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. MV60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 232 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. MV54 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Recital H. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Envy 50. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 246 υπέρ. Κατά αποχές Εμβε MV53 υπέρ κατά αποχές Εμβι MV55 υπέρ κατά αποχές Εμβι MV57 υπέρ κατά αποχές Εμβι MV59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμβη 61 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 245 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 248 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 249 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην τροπολογία 63 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στη συμβαστική 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε μία προσθήκη στην 17 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές, καθόλου σαφές. άρχεται η ψηφοφορία για την προσθήκη της Συμβαστικής 17. Κύριε Βίμ Βαντεκάμπ, ψηφίσαμε τη Συμβαστική 17 και τώρα ψηφίζουμε την προσθήκη της. Εντάξει. Σαφές. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται η προστίκη της συμβαστικής 17. Άρα περνάμε στην ξεχωριστή ψηφοφορία στην 272 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Επαληθεύουμε το δεύτερο τμήμα. Πέρας. 23-22. Άρα εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. 278 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 279 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 273 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 274 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 275 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 280 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Θέλετε παλήθευση της 280, γιατί 280 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 292 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 293 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 302 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται. Νομίζω, λέει η πρόεδρος. Θέλετε να επαληθεύσουμε. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία για την 302. Πέρας. Απορρίπτεται. 295 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 296. 296. Ε, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 19. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε μία προσθήκη στη συμβαστική 19. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 301 Υπέρ της 301. Παρακολουθείτε. Εντάξει, 301 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 307 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 334 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 303 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές άρχεται η ψηφοφορία 303 για την 303 Je ferme le vote. Πέρας εγκρίνεται 304 υπέρ. Κατά. Αποχές. 304 απορρίπτεται. 303 υπέρ. Κατά. Αποχές. 333 απορρίπτεται. 305 υπέρ. Κατά. Αποχές. 305 εγκρίνεται. 306 υπέρ κατά αποχές 306 εγκρίνεται 308 υπέρ κατά αποχές 308 απορρίπτεται 309 υπέρ κατά αποχές 309 εγκρίνεται. Να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. 309. Πέρας. Εγκρίνεται. 310. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 312 υπέρ κατά αποχές 312 εγκρίνεται και περνάμε κατευθείαν στην συμβιβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θέλετε να την επαληθεύσουμε αρχιετή ψηφοφορία Ναι, έχετε δίκιο. Απορρίπτεται. Περνάμε. Θα ψηφίσουμε λοιπόν. Την NV11. Το δεύτερο μέρος. Εντάξει. Υπέρ. Κύριε Ερτού, χαθήκατε. NV11. Το πρώτο μέρος δεν ψηφίζεται. Ψηφίζουμε το δεύτερο. Εντάξει. Υπέρ. Κατά. Προτιμώ να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 335. Μέχρι και την 342. Θα τις ψηφίσουμε όλες μαζί, εντάξει. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται όλες. Συνεχίζουμε. 345. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 345. Απορρίπτεται. Θέτε να την επαληθεύσουμε. Μάλιστα. Άρχεται η ψηφοφορία. 345. Πέρας. Αναπορρίπτεται. 346 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 348 υπέρ. Κατά. Αποχές. 348 εγκρίνεται 347 Α ναι 343 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές 347 κατέπεσε γιατί 348 εγκρίθηκε. Εντάξει. ...343 είμαστε τώρα, εντάξει. Δεν είναι σαφές λοιπόν, οπότε τίθεται σε ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 344 καταπίπτει. Τρακόσια πενήντα Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 349. Υπέρ. 349 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να την επαληθεύσουμε. 349. Πέρας. Απορρίπτεται η 349. 350 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 351 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 355 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 354 υπέρ κατά αποχές 354 εγκρίνεται. Τον υπότιλο ψηφίζουμε. Το υποκεφάλαιο υπέρ. Ε, κάπου χαθήκατε. Ναι, έχει ακόμα πολλές ψηφοφορίες. Ποιος είναι υπέρ του υποκεφαλαίου της Ανδύ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε απευθείας στην NV23 υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές. Α, την ψηφίσουμε λοιπόν την 23. Πέρας. Απορρίπτεται. 365 υπέρ κατά αποχές τι κάνετε 365 δεν ξέρω τι κάνετε ακριβώς Ωραία, είμαι αναγκασμένος να επαληθεύσουμε λοιπόν 365 αναγκασμένοι Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστικό 21β υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 369 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 370 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ΕΝΒΗ 26 μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 384 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Να ανταπαληθεύσουμε. 374. Πέρας. Απορρίπτεται. 375 υπέρ. Κατά. Αποχές 375 εγκρίνεται. 378 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 383 υπέρ. Κατά. Αποχές. 383 εγκρίνεται. 384 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην ένβη 28 δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπότιλος ένβη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ένβη 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές άνβη 32 μέρος δεύτερο εγκρίνεται 300 ε, Ναι, ναι. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Συμβαστική 22 εγκρίνεται. 390 υπέρ. Κατά. Αποχές. 390 εγκρίνεται. 391 υπέρ. Κατά. Αποχές. 391 εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. 23 εγκρίνεται. 401 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 402 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 403 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 404 υπέρ κατά αποχές 404 εγκρίνεται 405 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές 24 εγκρίνεται προσθήκη στην 24 υπέρ κατά υπέρ με συγχωρείτε κατά αποχές απορρίπτεται Περνάμε. Στην 419 ε, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 424 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και συνεχίζουμε. 446 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται το πρώτο μέρος. 444 υπέρ. Κατά. Κάποιος δεν ψηφίζει υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 447 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 448 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 442 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται υπό κεφάλαιο NV υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV μέρος δεύτερο 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε στην 462 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να την απολυθέψουμε. άρχεται η ψηφοφορία 462 Πέρας. Έχετε δίκιο. Εγκρίνεται. Τετρακόσια υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 466 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε τώρα στην NV42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 470 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 472 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να την επαληθεύσουμε να ψηφίσω κι εγώ Πέρας. 472 εγκρίνεται. 471 υπέρ. Κατά αποχές 471 εγκρίνεται. Περνάμε. 475 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 476 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 476 υπέρ κατά αποχές 478 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές θα ψηφίσουμε Άρχεται η ψηφοφορία. Ωραία. Ευχαριστώ, πέρας. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε. Συν 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Τροπολογία 4 εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. 5 εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε στην 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ένβη σκέψη 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV σκέψη 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, αιτιολογική σκέψη 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ναι ναι ωραία επερνάμε στην NVF υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NVG υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Να την επαληθεύσουμε μάλιστα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. AIDS. υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ανβι υπέρ. Κατά. Ε, ε, συγχωρείτε. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. 31 εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεν υπάρχουν άλλες. Για να περιμένετε. Α, ναι, ναι, ναι. EM. Συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τελική έκθεση. Πίστε ψηφοφορία. Άκρη ψηφοφορία. 25 υπέρ. Κατά. 10. 10 αποχές. Η έκθεση του κυρίου Άικχαουτ εγκρίνεται. Monsieur, écoute, vous voulez faire Κύριε Αικχάουτ θέλετε κάτι να μας πείτε, όχι Συνεχίζουμε. σε σχέση με την πρόταση απόφαση της κατεξιοδότηση πράξης, οδηγία 2010 κάθετος 40, τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 3, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ένα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πέντε υπέρ κατά απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το τελικό κείμενο. Πέρας. Εγκρίνεται 42 υπέρ με ομοφωνία. Ωραία, μπορούμε να προχωρήσουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν με την Ευρωμεσογειακή Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου σε σχέση με τις αεροπορικές υπηρεσίες. Ε, συγητής, ο κύριος Ρικέ. Τώρα είσαστε υπέρ ή κατά. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία. φαίνεστε κάπως χαμένοι εδώ στην πρώτη σειρά. Πέρας. Plus 44. 44 ομοφωνία. Συγχαρητήρια κύριε Ρικέ. Κύριε Μπας Εικχάουτ, θέλετε το λόγο, τον έχετε. Παρακαλώ να τον ακούσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να προτείνω την αναβολή αυτή τη ψηφοφορία. Πρώτα απ' όλα ε, προβλεπόταν ψηφοφορία μια ώρα και έχουμε ξεπεράσει αυτό το χρονικό διάστημα και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι αν ο κόσμο αρχίσει να φεύγει ε, δεν θα είναι ε, τόσο καλό και από δημοκρατικής άποψης. Δεύτερον, γνωρίζουμε ότι οι τροπολογίες αυτής της ε, έκθεσης είναι πολύ γενικές, πολλές θα απορριφθούν, οπότε δεν θα κρατήσει πολλή ώρα. Δεν ξέρω λοιπόν αν είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Και τρίτον, μπορούμε να το αναβάλουμε, παρόλο αυτό ο κόσμος πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ε, δεν θα είμαστε ε, στην ώρα μας για την ψηφοφορία της ΕΝΒΙ. Οπότε η ΕΝΒΙ θα ψηφίσει στις 23 Οκτωβρίου. εμείς μπορούμε να ψηφίσουμε πριν από αυτό. Παρ' όλα αυτά είμαστε ε, ε, ε, έγκαιροι όσον αφορά την Επιτροπή Ίντρα. Οπότε κάποια από τα ζητήματα που είναι κοντά στη δική μας Επιτροπή, όπως είναι τα βιοκαύσιμα, σε αυτά δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση και αυτό είναι το αρνητικό όμως δεδομένων όλων αυτών. Θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερο να μην ψηφίσουμε αυτή τη στιγμή. Είναι μια πρόταση και αν, θέλουμε να, αν οι υπόλοιποι θέλουν να συνεχίσουν τότε δεν έχω πρόβλημα, απλά θα κρατήσει αρκετή ε, ώρα. Alors, je vais demander les avis Λοιπόν, θέλω τη γνώμη σας. Κύριε Σαλίνη, τι λέτε. Η πρόταση ε, αναστολής είναι σωστή, γιατί η πρόταση είναι της Ήτρε και θα πρέπει να δώσουμε μία πολύ καλή εντολή στην ε, ΕΜΒΗ. Εγώ συμφωνώ να αναστείλουμε την ψηφοφορία. Ωραία. Η επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Ρεβονταλόν, κατανοώ ότι δεν μπορούν πολλοί να παραμείνουν για την ψηφοφορία, αλλά είναι πολύ κρίμα δεν μπορούμε όμως να υποστηρίξουμε τον εισηγητή, γιατί αν δεν ψηφίσουμε σήμερα, ό,τι σχετίζεται με την Επιτροπή ΕΜΒΗ δεν θα έχει αυτή τη συνδεσιμότητα. Και αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα. Κατανοώ ότι ορισμένοι βουλευτές πρέπει να εγκαταλείψουν την αίθουσα ή την εγκατέλειψαν ήδη. Έχουμε φυσικά πολύ φορτωμένη ημερήσια διάταξη. Πάντα έχουμε στην Επιτροπή μας. Μία διευκρίνηση. Εδώ μιλάμε για αποκλειστικά δικαιώματα της Επιτροπής Μεταφορών. Η κυρία Φώστερ τι λέει. Yeah, just a brief point. Ε, θα είμαι σύντομη ναι, και όλοι γνωρίζουμε ναι, ως ότι είναι δύσκολο ε, όταν προσπαθείς να τα προσθέσεις όλα αυτά σε ψηφοφορία όσον αφορά την πρώτη έκθεση του κυρίου Έκαρτ ήταν 40 σελίδες και πραγματικά δεν υπήρχαν αρκετές συμβιβαστικέ. Νομίζω ότι πρέπει να συστήνουμε όταν κάποιος έχει μια έκθεση πρωτοβουλίας ε, και την παρουσιάζει εδώ πέρα, τότε θα πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά, ούτως ώστε να υπάρχουν περισσότερες συμβιβαστικέ ε, και να έχουμε μια έκθεση η οποία να μην είναι τόσο ε, μεγάλη. Και όπως υπόθηκε πολύ σωστά, έχουμε αυτό το πράγμα ξανά. Δεν έχω πρόβλημα να μείνω εδώ να ψηφίσω. Όμως θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη μας ότι ο εισηγητές θα πρέπει να προσπαθεί ώστε να υπάρχουν συμφωνίες. Ε, δεν ξέρω ε, τι θα γίνει στο τέλος. Δεν έχω πρόβλημα να μείνω και να ψηφίσω αν θέλουν να συνεχίσουν και οι υπόλοιποι. Τι λένε οι φιλελεύθεροι. Madam Chair, I do understand. Ε, καταλαβαίνω τις ε, δυσκολίες ε, που αντιμετωπίζουν μερικές πολιτικές ομάδες όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας υπάρχουν και τα θετικά στο να ψηφίσουμε πριν από την ΕΝΒΗ λαμβάνοντας υπόψη μας ότι θα πρέπει να βρούμε ένα κενό στην Ολομελία του Στρασβούργου και να ψηφίσουμε εκεί. Allez, Madame Ayuto, Κυρία Γιούσο, α, κυρία Γιούτο μάλλον, δεν ε, καταλαβαίνω τη συλλογιστική ε, αναπομπής. Είχαμε προβλέψει ψηφοφορία για σήμερα το πρωί, δεν, έχει λόγο να, δεν έχουμε λόγο να διακόψουμε. Εάν βρούμε πολιτικούς λόγους, εντάξει, ας μην ψηφίσουμε αλλά είναι πολύ αδύναμο αυτό το επιχείρημα που προέβαλε ο κύριος Eichhout. Δεν έχω τη γνώμη της Γκούε. Παρακαλώ. speaking speaking. Ε, θα πρέπει να αρχίσουμε να ψηφίζουμε και να ε, πάμε σπίτι. Αυτό δεν είναι σωστό. Ποιος είναι η υπέρ της αναστολής της ψηφοφορίας αναστολή της ψηφοφορίας της έκθεσης. Κατά. Ε, ε, ε, Ήταν σαφές το αποτέλεσμα ποιοι θέλετε να ψηφίσουμε σήμερα. Ποιος λέει ναι για τη σημερινή ψηφοφορία. Κατά. Η πλειοψηφία λέει όχι. Άρα δεν ψηφίζουμε την έκθεση Bas Άικχαουτ. Κύριε Άικχαουτ θα ήθελα να έρθετε εδώ στα έδρανα της Γραμματείας για να βρούμε μία ημερομηνία. Τέλιτσκα. Θα κάνουμε μία δεύτερη ψηφοφορία με την πρόταση την οποία έγινε ότι θα ψηφίσουμε πριν την ψηφοφορία της ΕΝΒΗ. Καταλαβαίνω ότι τη Δευτέρα το απόγευμα υπάρχει μία ψηφοφορία της ΕΝΒΗ, όμως γίνεται να ψηφίσουμε πριν από αυτό. Ε, είναι πολύ λογικό να έχουμε μία ψηφοφορία πριν ε, την ε, γνωμοδότηση της ΕΝΒΗ. Όταν μιλά ένας συνάδελφος, τον σεβόμαστε. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Τέλιτσκα, παρακαλώ. Παρακαλώ λίγο σεβασμός για τους συναδέλφους. Κύριε Τελίτσκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, ε, πιστεύω ότι θα είχαμε μια ψηφοφορία και για αυτό το οποίο ε, πρότεινα ότι θα ψηφίσουμε πριν από την ε, ψηφοφορία της ΕΝΒΗ. Καταλαβαίνω ότι είναι η ψηφοφορία το βράδυ, το απόγευμα της Δευτέρας, όμως καλώ όλους τους συναδέλφους και πολιτικές ομάδες να ψηφίσουμε πριν από την ΕΝΒΗ. Δάλλως θα ήταν λάθος και σίγουρα θα ε, ε, δυσχεραίναμε τη θέση την οποία θέλουμε να λάβουμε. Πιστεύω αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε τώρα είναι ότι είναι μια καλή πρόταση. Ε, το, χρονοδιά, το χρονοδιάγραμμα είναι περιορισμένο, οπότε δεν μπορούμε να αποφασίσουμε αμέσω. Όμω θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό. Όμω θα είναι περιορισμένε οι δυνατότητε, διότι Δευτέρα απόγευμα ψηφίζει η ΕΝΒΗ, Δεν ξέρω τι ώρα ακριβώ, όμω ίσω υπάρχει δυνατότητα να το κάνουμε λίγο πιο πριν. Οπότε θα πρότεινα τη, ε, τη θέση του κυρίου Ντελίκα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να λειτουργήσει το planning, αλλά μπορούμε να, το, ε, να βρούμε μια λύση. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ψηφίσουμε την έκθεσή σας πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Γιατί λέτε Ήτρε. Α, γιατί επί της ουσίας ε, γνωμοδοτεί Ήτρε. Κύριε Μπάς Άικχαουτ, παρακαλώ ελάτε εδώ στη γραμματεία για να δούμε πότε θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε την έκθεσή σας. Ωραία, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με τη συνεδρίασή μας. Ceux qui veulent quitter la salle le font en silence, s'il vous plaît. Παρακαλώ να αποχωρήσετε ήσυχα όσοι αποχωρείτε. Συνεχίζουμε με μια ανταλλαγή απόψεων με τη Γενική Διεύθυνση MOVE σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα ως προς δύο πτυχές. Εσωτερική αγορά και κοινωνικός τομέας. Παρακαλώ Όσοι θέλετε αποχωρήστε, αλλά ήσυχα, χωρίς να ενοχλείτε. Voilà, c'est mieux. Ωραία, καλύτερα τώρα. Όπως γνωρίζετε, η Επίτροπος Βιολέτα Μπούλτς ε, παρουσίασε το πρόγραμμα στις 31 Μαΐου και στην Επιτροπή Μεταφορών στις 19 Ιουνίου. Σήμερα έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων με τη Γενική Διεύθυνση MOVE μετά θα έρθουμε σε διαβούλευση με τους εμπειρογνώμονες κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης με την Επιτροπή Απασχόλησης στις 16 Οκτωβρίου και κατά την ακρόαση στις 22-23 Νοεμβρίου. Αυτές οι συζητήσεις θα βοηθούσαν τους εισηγητές να προετοιμάσουν ε, τα σχέδια γνωμοδότησης για τον Ιανουάριο προτείνω να διαχωρίσουμε τη συζήτηση σε δύο τμήματα, να αρχίσουμε με τις κοινωνικές πτυχές και τις πτυχές αγοράς και να μετά να μιλήσουμε για τα οδικά τέλη. Γι' αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Βέρνερ. Είναι εδώ η κυρία Βέρνερ. Καλημέρα σας κυρία Βέρνερ. Θέλετε να έρθετε να καθίσετε εδώ. Α, προτιμάτε να μείνετε εκεί που είστε. Εντάξει από τη Γενική Διεύθυνση MOVE για να μας ε, παρουσιάσει την κατάσταση της αγοράς ως προς την κοινωνική πτωχή, δηλαδή την πρόσβαση στην αγορά και στα επαγγέλματα σε σχέση με τους οδηγούς ε, ιδιαίτερα των αυλωμένων οχημάτων. Έχετε 10 λεπτά και μετά θα λάβουν το λόγο οι και οι σκιώδεις και θα δώσω το λόγο στη συνέχεια σε όσους τον επιθυμούν. Πρόκειται για ένα θέμα πολύ πολιτικοποιημένο. Νομίζω ότι πολλοί θα θέλουν να λάβουν το λόγο. Θα ήθελα να σηκώσω το χέρι για να ξέρω ποιοι θέλετε να μιλήσετε και θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε στη διάθεσή μας κάτι λιγότερο από δύο ώρες για αυτή την ανταλλαγή απόψεων για τα νομοθετικές προτάσεις. Θα ήθελα λοιπόν να περιοριστείτε στις παρεμβάσεις έτσι ώστε να έχουμε απαντήσεις. Δίνω το λόγο στην κυρία Βέρνερ για να μας παρουσιάσει για 10 λεπτά τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτή την πτυχή του θέματος. Έχετε το λόγο. Euh, Ευχαριστώ. Είμαι πολύ καλά εδώ γιατί ε, πλαισιώνουμε από όλους τους ε, συναδέλφους, διότι σήμερα θα θέλαμε να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας λεπτομερώς. Στις 31 ε, Μαΐου λοιπόν έχουμε ένα ευρύτερο ε, πακέτο σχετικά με την ε, Ευρώπη σε κίνηση, η διασυνδεδεμένη κινητικότητα και αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει η Κομισιόν σε αυτό το πλαίσιο είναι να ακολουθήσει μια γενικότερη προσέγγιση σε ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τις οδικές μεταφορές. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι υπάρχουν αρκετές προκλήσεις και συμβαίνουν αρκετές αλλαγές λόγω των νέων τεχνολογιών και των νέων επιχειρηματικών μοντέλων που κάνουν την κινητικότητα πιο βιώσιμη, ταυτόχρονα όμως έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και νέε ανισότητε. Γι' αυτό το λόγο είναι προ ε, προς το συμφέρον μας να εξετάσουμε τις προκλήσεις και τα ε, επιχειρηματικά μοντέλα. Η κινητικότητα ε, βιώνει τρομερές αλλαγέ ε, και αυτό γίνεται και στο πλαίσιο της δέσμευσή μα να επιτύχουμε τους κλιματικούς στόχου και να έχουμε έναν δίκαιο τομέα. Επίσης, οι προτάσει αυτές έχουν μια ισορροπημένη προσέγγιση και συνδέονται στενά με την, με την, με την πλευρά της ε, αγοράς ε, στο οποίο θα επικεντρωθούμε στον πρώτο κύριο διαλόγου σήμερα. Ο στόχος λοιπόν είναι να προωθήσουμε μια αποτελεσματική και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά διασφαλίζοντας επίσης ε, δίκες, δίκες συνθήκες εργασίες για τους οδικούς μεταφορείς και επίσης έχουμε και περιβαλλοντικό περιβαλλοντικούς ε, στόχους ε, και αυτό σχετίζεται με τη χρήση των υποδομών αλλά και ε, να εισάγουμε την ψηφιοποίηση στον τομέα το οποίο θα συζητήσουμε στο δεύτερο γύρο. Τώρα όσον αφορά την εσωτερική αγορά γνωρίζουμε ότι έχουμε σοβαρά ζητήματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Δεν λειτουργεί τόσο καλά όσο θα θέλαμε αυτή τη στιγμή. Ε, θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερες προτάσεις που θα υιοθετηθούν πριν από ε, τις ευρωεκλογέ ε, το 2019 και γι' αυτό το λόγο θα θέλουμε να επιταχυνθεί όλη η διαδικασία. Επίσης, πριν περάσω στην ουσία θα ήθελα να αναφέρω και μία άλλη σειρά πρωτοβουλειών το δεύτερο πακέτο κινητικότητας το οποίο θα προσθεθεί στην ημερήσια διάταξη στις 8 Νοεμβρίου στην Κομισιόν. Έχουμε μια ε, δευτερεύουσα νομοθετική πρόταση ε, που αφορά την οδηγία ε, καθαρών οχημάτων. Έχουμε την πρόσβαση στην αγορά πούλμαν και λεωφορείων και εκεί υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες. Έχουμε την αξιολόγηση και το σχέδιο δράσης σχετικά με τα εναλλακτικά καύσιμα ε, και, τη χρήση περισσότερων υποδομών ε, φορτισής. Ε, έχουμε νομοθεσίες σχετικά με τα πρότυπα για την φόρτιση οχημάτων και υποδομές αυτών και επίσης έχουμε την συνδυαστική οδηγία μεταφορών που συνδέεται και με την οδηγία καμποτάζ. Ε, τώρα κάποια ε, βασικά χαρακτηριστικά της πρότασης ε, θα είμαστε σύντομοι. Όσον αφορά το κομποτάζ, η πρόταση είναι η απλοποίηση των κανονισμών ούτως ώστε να εφαρμόζονται πιο εύκολα. Στόχος είναι όχι μόνο να ανοίξουμε ή να κλείσουμε την αγορά. Έχουμε εξετάσει προσεκτικά ούτως ώστε να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Είδατε την αξιολόγηση, στην αξιολόγηση αντικτύπου μας. Επίσης έχουμε το θέμα των εικονικών εταιριών όπου ε, στόχος είναι η ενίσχυση των ε, κριτηρίων ε, για να μπορούν να λειτουργούν τέτοιες εταιρείες σε συγκεκριμένες χώρες και επίσης θέλουμε διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ούτως ώστε να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι. Επίσης, όσον αφορά τα εμπορικά οχήματα, τα μικρότερα βαν, εδώ επεκτείνουμε το εύρος των κανονισμών για την πρόσβαση σε διάφορους επαγγελματίες. Προσπαθούμε ε, να ε, μην κάνουμε πολύπλοκη την νομοθεσία, παρόλα αυτά να υπάρχει ένα ε, κάποιο επίπεδο επαγγελματοποίησης, διότι υπήρξε μεγάλη διαμαρτυρία για το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται βαν για να παρακαυθούν οι κανονισμοί για τα βαρέα οχήματα. Επίσης, έχουμε την ε, πρόταση να επεκτείνουμε ε, την ε, ευελιξία για την ενοικίαση αυτοκινήτων κάτι το οποίο θα επέτρεπε την προσαρμογή με βάση τις εποχιακές ανάγκες. Ε, για να ε, έχουμε τις απαραίτητες συνθήκες εργασίας ξεκαθαρίζουμε ότι οι οδηγοί θα πρέπει να ε, σέβονται τις, τους κανονισμούς διαλύματος και ξεκούρασης αυτό συζητάται ήδη στο Συμβούλιο και έχουν προχωρήσει αρκετά και θα πρέπει να εξετάσουμε επίσης τα πάρκινγκ ως ένα κομμάτι της λύσης. Ε, κάναμε μία έρευνα πάνω σε αυτό ε, για να γίνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα ε, και υπάρχουν τα χρήματα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2017 και ο χρόνος είναι πολύ καλός. Επίσης έγιναν προτάσεις για να αλλάξουμε τις εβδομαδιαίες περιόδους διαλύματος για τους οδηγούς και την ανάγκη να επιστρέψουν στο σπίτι. Αυτό έχει ως στόχο να, να βοηθήσει την ευελιξία ούτως ώστε οι να κανονίζουν τα ταξίδια τους και ταυτόχρονα να βελτιώσει τι συνθήκε εργασία, αλλά και την ισορροπία εργασία και προσωπική ζωής ε, συνεισφέροντα την οδική ασφάλεια και ταυτόχρονα κάνοντας το επάγγελμα πιο ελκυστικό. Γνωρίζουμε ότι σε κάποιες χώρες υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. Επίσης ε, προτείνουμε συνθήκε για την εφαρμογή ε, των κανονισμών του οδηγίας περί αποσπάσεως εργαζομένων ε, στην Επιτροπή δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συγκεκριμένη οδηγία μπορεί να εφαρμοστεί στις οδικές μεταφορές και προτείνουμε ένα καθεστώς το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του ε, με ε, ελάχιστες διοικητικές απαιτήσεις. Τέλος, θέλουμε να προτείνουμε την εναρμόνιση της εφαρμογής και να ενισχύσουμε ε, την ε, διοικητική συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ενθαρρύνουμε τη χρήση και την ανάπτυξη ψηφιακών εγγράφων τα οποία θα μειώσουν το διοικητικό κόστος ε, ε, για τους ελέγχους και την εφαρμογή. Είναι πολύ σημαντικό ε, με βάση τους αριθμούς οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί όσον αφορά το διοικητικό άχθος ε, το οποίο ανέρχεται στα 3 με 5 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 15 χρόνια. Τώρα όσον αφορά τη διαδικασία όπως ε, θυμάστε προτάθηκε στην, στην Ολομέλεια ε, η θέση την ημέρα που υιοθετήθηκε από την Κομισιόν. Επίσης είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε ερωτήματα στο Γενικό ε, Διευθυντή και είχαμε την δυνατότητα να συναντηθούμε με τους γνωμοδότες και να παρουσιάσουμε τις προτάσεις βρισκόμαστε σε καθημερινή επαφή με το Κοινοβούλιο σε διάφορα επίπεδα για να μπορέσουμε να απαντήσουμε όλα τα ερωτήματα. Ε, τώρα προς το Συμβούλιο ε, θα ήθελα να ε, χαιρετήσω την Εστονική Προεδρία που έχει εργαστεί άμεσα και γρήγορα πάνω σε αυτό και έχει κάνει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά την εσωτερική αγορά και τον κοινωνικό τομέα και ε, το ε, Συμβούλιο στην ε, συνάντηση της Τη 5 η Δεκεμβρίου θα συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω, θεωρούμε ότι αυτό ε, θα ανοίξει την, ε, θα δώσει τη δυνατότητα ούτω ώστε να ψηφιστεί κατά τη Βουλγαρική ε, Προεδρία και στη συνέχεια θα μπορέσουν να ακολουθήσουν οι τριμερεί διάλογοι. Η Προεδρία επίσης σκοπεύει στη Σύνοδο του Δεκεμβρίου να συζητήσει και το ζήτημα των οδικών τελών. Ε, ήδη βλέπουμε κάποιες ε, συμβιβαστικές λύσεις από την πλευρά των καλών κρατών μελών όπως σε διάφορα σημεία όπως είναι για παραδείγμα ε, το ζήτημα των εικονικών εταιριών όπως επίσης και για τα ελαφρά εμπορικά οχήματα για την καλύτερη χρήση του ταχόγραφου ε, για την εφαρμογή νομοθεσία συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Ε, επίσης υπάρχουν άλλα θέματα όπως είναι το καποτάζ, ε, τα οποία ε, για τα οποία επίσης θα υπάρχουν συζητήσεις ε, όμως υπάρχει μια επικοδομητική ατμόσφαιρα και ήδη μπορούμε να δούμε ότι θα βρούμε κάποιες ε, λύσεις για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του συστηματικού καμποτάζ και όσον αφορά τις κοινωνικές προτάσεις και εκεί έχουμε βρει κοινό έδαφος όπως είναι για παράδειγμα τη διανυκτέρευση σε καμπίνες και την επιστροφή στο σπίτι. Όσον αφορά τους, τα κοινωνικά ζητήματα επικεντρωνόμαστε στις συζητήσεις ε, για την ε, γενική οδηγία ε, περί αποσπάσεως εργαζομένων το οποίο θα γίνει τέλη Οκτωβρίου και είχαμε μία συζήτηση χθες όπου έχουμε δύο στρατόπεδα από τα κράτη-μέλη Χαίρομαι λοιπόν που, ε, που βρισκόμαστε εδώ και ε, είστε τόσοι πολλοί ε, για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και θα συνεργαστούμε και με τις Επιτροπές Απασχόλησης και Περιβάλλοντος για να έχουμε έναν επικοδομητικό διάλογο. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι στόχος για την Κομισιόν είναι να υιοθετήσουμε ως το δυνατόν περισσότερες προτάσεις ε, πριν από αυτή τη θητεία του Κοινοβουλίου ε, είδατε ότι ο, ε, ο κύριος Γιούνκερ κάλεσε να γίνει μια γρήγορη οθότηση αυτού του πακέτου. Ο χρόνος μας πιέζει και είμαστε εδώ για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και θα χαρούμε επίσης να πάρουμε και ερωτήματα και να σας τα απαντήσουμε γραπτό σε περίπτωση που δεν μας επιτρέψει ο χρόνος να απαντήσουμε σε όλα. Ευχαριστούμε πολύ την Επιτροπή για αυτή την παρουσίαση που είναι εκτενής. Φυσικά χρειάζεται και περαιτέρω εμβάθυνση. Θα δώσω το λόγο στους εγγεγραμμένους και αρχίζω με τον κύριο Ντεγκράντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω ε, μία ε, παρέμβαση σε σχέση με ιστορικά δεδομένα. Το σύνταγμα της Ισπανίας ισχύει από το 1978, το νέο, ε, το νέο σύνταγμα, από το οποίο ευεργετούνται όλοι. Και το ίδιο αφορά και την Επιτροπή μας, η οποία ε, διέπεται από μία ένομη τάξη. Μιλάμε για ένα πιο ολοκληρωμένο και διατροπικό σύστημα μεταφορών, καλύτερες συνθήκες εργασίες, μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η απότεροι στόχοι, οι οποίοι είναι ε, πενετέοι. Υποστηρίζουμε την ε, εβδομαδιαία ε, ανάπαυση, το χρόνο ανάπαυσης, όπως προβλέπεται από τον Κομισιόν, αλλά ε, υπάρχουν πολλές αμφιβολίες και αμφισημίες, όπως είπε και η κυρία Βέρνερ, δηλαδή θα πρέπει να μπορούν να αναπαύονται σε κατάλληλους χώρους και όχι μέσα στα οχήματά τους. Επίσης θα πρέπει να μιλήσουμε και για επιθεωρήσεις, διότι πολλές φορές τα οχήματα δεν είναι ιδιαίτερα εξυγχρονισμένα. Ως προς την απόσπαση εργαζομένων θα πρέπει να προσαρμοστούμε στην ε, πραγματικότητα, γιατί τα μέτρα δεν είναι αναλογικά. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε ολιστικά με το θέμα της απόσπασης ε, των εργαζομένων, γιατί δυστυχώς δεν είναι αναλογικά αυτά τα μέτρα. Επίσης, η πρόσβαση στην αγορά αλλάζει το κατόφλι σε σχέση με την πρόσβαση των ε, μικρών οχημάτων, δηλαδή κάτω από τους 3,5 ε, 3,5 τόνους. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να ε, βρεθεί μία κατάλληλη και αναλογική λύση. Θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε στην Επιτροπή ότι όλες αυτές οι συνδυασμένες προτάσεις στην ουσία οδηγούν σε ε, νικητές και ιτημένους. Δηλαδή κερδίζουν τα κράτη που βρίσκονται στο κέντρο της Ευρώπης και χάνει η περιφέρεια. Γι' αυτό θα πρέπει να μην υπάρχει αυτή η ασυμμετρία στις μεταφορές, ιδιαίτερα όσον αφορά τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Νίλσεν έχει το λόγο. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Θα προτιμήσω ε, να ε, επαναλάβω τα λόγια του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γιούνκερ, ο οποίος επανειλημμένως είπε ότι ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να έχουμε κοινωνικό ντάμπινγκ και αυτό είναι μια καλή αρχή. Όταν εργαζόμαστε πάνω σε ένα τέτοιο θέμα Και γι' αυτό το λόγο με ενοχλεί όταν μιλάμε για επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία αποσκοπούν στο να κάνουμε ένα shopping κανόνων από τις διάφορες χώρες. Έτσι λοιπόν μπορείς να ιδρύσεις μια εταιρεία σε μια χώρα όπου έχει χαμηλότερους φόρους ή χαμηλότερα κόστη. Αυτό είναι κοινωνικό dumping και θα πρέπει να εργαστούμε κατά αυτού. Βλέπω αρκετές εικονικές εταιρείε και το πώς ε, σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ε, ο κανονισμός μπορεί να γίνει ε, καλύτερος. Τώρα από την άλλη όσον αφορά τα διαλύματα δεν είναι το θέμα αν θα είναι 7, 5 ή 2 ημέρες. Το πιο σημαντικό είναι μπορείς ε, να ε, το ελέγξεις, να το παρακολουθήσεις όλο αυτό αν εφαρμόζεται. Η Κομισιόν προτείνει τα κράτη-μέλη να φέρουν την ευθύνη για αυτό. Και βέβαια το υποστηρίζουμε αυτό, ε, θα πρέπει να είναι δυνατό να γίνει αυτό έχουμε ε, τους ταχόγραφους ε, στα οχήματα οι οποίοι, οι οποίοι θα λειτουργούν σωστά και έτσι λοιπόν θα είναι πιο εύκολο να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε και επίσης ε, θα ήταν πιο εύκολο να κάνουμε κάτι εναντίον αυτών που παραβιάζουν τους κανόνες. Ε, τώρα το ζήτημα του καποτάζ είναι ένα θέμα το οποίο επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, πρέπει να ε, κάνουμε κάτι γι' αυτό αν θέλουμε να ακολουθήσουμε και να τηρήσουμε την πρόκληση του ε, κυρίου Γιούγκερ. Τώρα όσον αφορά την οδηγία μου αρέσουν οι συνδυαστικές λύσεις, λύσεις μεταφορές και στις διάφορες περιοχές περιοχές ε, της Ευρώπης μπορούμε να βρούμε ε, καλές πρακτικές όμως ε, το λύνει αυτό η αγορά από μόνη της θα έχουμε ένα μια συνδυαστική οδηγία όμως θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί για να παρακαμφθούν οι κανόνες του καποτάζ και τέλος η... ο έλεγχος και η παρακολούθηση αυτό είναι το πιο σημαντικό Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος ε, Ζήλε έχει το λόγο. Well, uh, I think it's, uh, Δεν υπάρχουν πολλοί στην αίθουσα. Θα ήθελα όμως να πω λίγα λόγια. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ την Κομισιόν για τις εξηγήσει. Ε, δεν ξέρω αν ξέρετε πότε θα ετοιμάσει το Συμβούλιο αυτό το θέμα. Μας ενδιαφέρει. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε τόσο μεγάλες ε, διαφορές ε, κάποια κοινωνικά ζητήματα, αλλά από ό,τι φαίνεται στο Συμβούλιο θα έχουμε δύο μπλοκ κρατών και εδώ μέσα μάλλον θα έχουμε δύο μπλοκ ευρωβουλευτών. Αυτό φαίνεται ότι είναι το, το πρόβλημα. Ο μακροπρόθεσμος στόχος μου βεβαίως δεν έχει σχέση με το πακέτο αυτό, είναι να αν μιλάμε για ενιαία αγορά ο ορισμός του καμποτάζ είναι λάθος. Μιλάμε για μία ενιαία αγορά ή για 28 αγορές ε, και για κοινωνικές συνθήκες. Εντάξει, ίσως μπορούμε να ορίσουμε κάποιου ελάχιστους κοινωνικούς όρους ε, και μετά να ανταγωνιστούμε. Αυτό είναι το, το Δεν θα επιτύχουμε με αυτήν την φιλοσοφία ε, στη συζήτηση αυτή. Απλά θα ήθελα να πω από τους συναδέλφους, στους συναδέλφους ότι πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι είμαστε διχασμένοι ως ε, προς αυτό όσον αφορά την αγορά των οδικών μεταφορών. Π.χ. επιστρέφοντας στη, ε, στη χώρα του, στην πατρίδα του. Ε, τι είναι η, η χώρα αυτή. Είναι η υπηκότητα του οδηγού, είναι η πινακίδα του αυτοκινήτου, τι από όλα αυτά και γιατί οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν ε, στον ελεύθερο χρόνο του να πάει, σε, να πάει κάπου αλλού που να μην είναι η χώρα υπηκότητας και διαβατηρίου. Περίεργη έννοια και δεν έχω ακόμα λάβει κάποια απάντηση από αυτούς που προετοίμασαν την πρόταση. σου στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου υπάρχει μια πιο ξεκαθαρή κατάσταση. Α, δεν έχω ακούσει μια σαφή απάντηση επί του θέματος. Αυτά για την ώρα. Και να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν συμβασμό. Και κάτι άλλο. Μου είπαν ότι η Επιτροπή απασχόλησης ετοιμάζει μόνο εκτιμώντας. Ε, ξέρετε, αν πάει στην Ολομέλεια έτσι, ε, τα εκτιμώντας δεν είναι διατακτικό δεν είναι, δεν είναι κάποια νομική διάταξη. Τα μπερδεύουμε όλα μαζί γιατί βεβαίως θα μας απασχολήσει εδώ και καιρό και στην καλύτερη περίπτωση θα το ολοκληρώσουμε στο τέλος της θητείας. Ε, και μεταξύ δεν υπάρχει νομική βεβαιότητα. γιατί υπάρχει βεβαίω μεγάλη πίεση για την οδηγία περί αποσπασμένων εργαζομένων από κάποιους αρχηγούς κρατών, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουν αυτές οι αβεβαιότητες, γιατί αυτή τη στιγμή είναι, υπάρχουν μόνο κάτι εκτιμώντας στην σχετική οδηγία. Σας ευχαριστώ κύριε Τζίλε. ο Τελίνσκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, έχουμε ένα από τα πιο σημαντικά νομοθετήματα εδώ πέρα μπροστά μας. είναι πολιτικά ευαίσθητο, είναι τεχνικό, έχει πολλές συνέπειες, μιλάμε για την αγορά και την κοινωνική διάσταση. Και ξέρουμε ότι έχουμε αποκλίνουσες απόψεις και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Και ταυτόχρονα, ενώ δεν έχουμε ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις στην Επιτροπή ή τις Επιτροπές. Έχουμε κράτη-μέλη τα οποία λαμβάνουν ε, μεμονωμένα μέτρα, τα οποία μπορεί να θεωρηθούν ως κάτι το προσωρινό, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι επηρεάζει και τις θέσεις των ε, κρατών μελών και το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω έκκληση θα ήθελα η Κομισιόν να είναι σε επαφή με τα κράτη-μέλη που έχουν λάβει ή θα λάβουν μονομερή νομοθετικά ή μη νομοθετικά μέτρα και να τους ζητήσει να μπουν κατά μέρος για να υπάρξει κάποια ποιοτική νομοθεσία. Δεύτερον, ναι, μιλάμε για κοινωνικό ντάμπινγκ, εσωτερική αγορά Ο καθένα καταλαβαίνει κάτι διαφορετικό με αυτέ τι λέξεις βεβαίω, ε, όταν λέμε κοινωνικό dumping ε, και ίσως και με τις λέξεις εσωτερική αγορά. Λοιπόν, πρέπει να ε, επιτύχουμε. Αν είναι να επιτύχουμε και αν θέλουμε ένα προβλέψιμο και δίκαιο νομικό πλαίσιο, θα πρέπει κάθε πολιτική ομάδα να αναζητήσει συμβιβασμό. Αλλιώ θα έχουμε ένα μακροσκελέστατο κατάλογο ψηφοφοριών με πολλές τροπολογίες και θα προκύψει ένα υβρίδιο. Απευθύνω λοιπόν έκκληση σε όλους. Σαφώς υπάρχει και προστατευτισμός, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις, ας το παραδεχτούμε, όπου το φορτηγό μια εταιρεία μπορεί να μην είναι καν από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, μπορεί να είναι από αλλά μπορεί να είναι και από μια γαλλική, ολλανδική εταιρεία, ε, φορτηγά τα οποία διατρέχουν κάποια κράτη-μέλη, όχι μόνο δυτικοευρωπαϊκά, επί εβδομάδες και ο οδηγός ε, κοιμάται κάπου σε πάρκινγκ και αλλού. Αυτό είναι το ένα άκρο. Το άλλο άκρο είναι να μπούμε στον πειρασμό να διαταράξουμε την εσωτερική αγορά και κάποιοι από εμά, κάποια κράτη-μέλη, έχουν αυτήν την φιλοδοξία. Και τα δύο είναι επικίνδυνα και θα έχουν επιπτώσεις όχι μόνο στις μεταφορές αλλά και σε άλλα οικονομικά συμφέροντα και στην ανάπτυξη σε κάποια άλλα σημεία τώρα. Ναι, σαφώς ε, πρέπει να αλλάξει κάπως ο χρόνος ανάπαυσης, αλλά αυτό το οποίο προτείνεται πάλι είναι με κάποιες ασαφείς διατάξεις ε, και ορισμούς που δεν ε, ε, έχουν βεβαίως πάντα σοβαρές ε, μελέτες επιπτώσεων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στο τέλος της περίοδου α, λέει, θα επιστρέψει ο οδηγός αλλά όχι το φορτηγό. Ε, το θέμα είναι το φορτηγό και όχι ο οδηγός. Δηλαδή αν ε, υπήρχα εγώ επιχείρηση μπορούσα εύκολα, ευκολότατα να φέρω τον οδηγό σε κάποιες ώρες με το Flexibus π.χ. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν τα πάρκινγκ. Τα, κυρία Πρόεδρε δεν ξέρω. Ε, τελειώνει ο χρόνος, το ξέρω, αλλά είτε κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση στο πακέτο κινητικότητας ή θα κάνουμε κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Ε, εγώ θέλω μια σοβαρή συζήτηση. να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το καμποτάζ. Κόβουμε π.χ. τον αριθμό ημερών ή τα πρόστιμα ή τις θέσεις παρκαρίσματος. Το πακέτο είναι καλό πακέτο με πολλά όμως προβληματικά σημεία. Απευθύνω έκκληση λοιπόν να έχουμε το πολιτικό θάρρο να αντισταθούμε στις πιέσεις που υπάρχουν ε, και στις δύο πλευρές, να βγάλουμε ένα καλό πακέτο και για, την, για τις μεταφορές και για τη βιομηχανία μας. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Θα κατεβάσω κάποιες προτάσεις για το δικό μου το θέμα, αλλά ας είμαστε λογικοί και υπεύθυνοι. Ευχαριστούμε κύριε Τελίτσκα. Και εγώ θα λάβω το λόγο ως συνεισηγήτρια. Επιτέλους, θα έχουμε ένα πακέτο για την κινητικότητα, όπου αυτή η κοινωνική πτυχή δεν θα μας επιτρέψει να λέμε ότι δεν υφίσταται πρόβλημα. Υπάρχει και πρέπει να βρεθούν λύσεις. Όλοι μιλήσαν για κοινωνικό dumping. Αυτό είναι το δηλητήριο του ευρωπαϊκού προγράμματος. Γι' αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε κοινωνικά. Δεν θέλουμε να θέσουμε τους εργαζόμενους τους μεν κατά τον δε από πλευράς ανταγωνισμού. Θέλουμε να τους προστατεύσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνολικά. Αυτό είναι ο απότερος στόχος. Η Επιτροπή μας λέει ότι τελείωσαν οι εικονικές επιχειρήσεις. Όλοι συμφωνούμε ότι ναι. Επιτέλους. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει το πρόβλημα μέχρι το 2017. Άρα θα τις αντιμετωπίσουμε. Και ε, αν ορισμένε επιχειρήσεις άνοιξαν ψευδοθυγατρικές, σε άλλα κράτη-μέλη τα θύματα είναι πάντα τα ίδια. Οι μισθωτοί, τους οποίους εκμεταλλευόμαστε με χαμηλούς μισθούς και με συνθήκες εργασίας οι οποίες είναι απαράδεκτες. Το θέμα είναι πρώτης τάξης Μιλάμε για έλεγχο, για επιθεωρήσεις. Άρα θα πρέπει να μιλήσουμε για κυρώσεις, κάτι το οποίο δεν ακούω. Υπάρχουν επιχειρήσεις ακόμα και εδώ στο Βέλγιο που μεταχειρίζονται κατά αυτόν τον τρόπο τους εργαζόμενους. Γι' αυτό θα πρέπει να αρχίσουν οι κυρώσεις. Δεύτερα, ως προς το καμποτάζ. Αυτή τη στιγμή επιτρέπεται το καμποτάζ με βάση ένα διεθνές ε, δρομολόγιο προς την χώρα υποδοχής του καμποτάζ. Και δεν καταλαβαίνω γιατί η Επιτροπή θέλει να μειώσουμε την αδειοδότηση στις πέντε ημέρες. Και αυτό γιατί σας το λέω. Γιατί αν στις πέντε μέρες τα φορτηγά κάνουν αυτά τα δρομολόγια, έτσι τα απελευθερώνουμε. Και εδώ μιλάμε για συνθήκες εργασίας και για οδική ασφάλεια. Τη στιγμή που ο οδηγός πρέπει να πάει γρήγορα, πολύ γρήγορα, για να εκπληρώσει την αποστολή του, τάχιστα, δεν υπάρχει οδική ασφάλεια. Άρα να μου εξηγήσετε γιατί σήμερα υπάρχει αυτός ο περιορισμός και γιατί έρονται τα περιθώρια και τα όρια. Εντάξει για τους ταχογράφους, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Είτε θα έχετε ε, ταχογράφους από το 2020 όταν βγούμε από τις ε, διαπραγματεύσεις δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό ισχύει και για τους ελέγχους. Δεν θα πρέπει να μιλάμε μόνο για τεχνολογία. Θα πρέπει να προχωρήσουμε. Και εγώ υπερεύει το χρόνο μου. Γιατί να μην έχουμε έναν ευρωπαϊκό οργανισμό ελέγχων με ευρωπαίους ε, επιθεωρητές. Πριν είχαμε τελωνιακούς. Γιατί να μην έχουμε επιθεωρητές ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα είχαμε τη δυνατότητα. Ε, μίλησα για ευρωπαϊκό σώμα επιθεωρητών και όχι για οργανισμό. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Λούγκριλ. Tack för det. Till skillnad från medlemmarna i GD Move och de flesta av mina kollegor här inne så har jag ju tillbringat όπως ε, είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοί μου, ε, αντιμετωπίζουμε ε, την προσωπική ζωή, την επαγγελματική ζωή από το 1994 οδηγό φορτηγά και ξέρω πώς λειτουργεί η αγορά στη χώρα μου, το έχω βιώσει μέχρι και το 1995 οπότε και η Σουηδία δυστυχώς αποφάσισε να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαι απογοητευμένος διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ενισχύσει καθόλου την ανταγωνιστικότητα αντιθέτως οι κανονισμοί έχουν καταστρέψει την ανταγωνιστικότητα επιτρέποντας ε, φορτηγά από ε, χαμηλόμιστες χώρες ε, με οδηγούς σκλάβους να ανταγωνιστούν σοβαρές εταιρείες που παίρνουν χρήματα για να πληρώσουν φόρους και κοινωνικές συνοσφορές κάτι το οποίο αποτελεί τη βάση της κοινωνικής πρόνοιας μιας χώρας και τώρα μιλάμε για το καποτάζ ε, το οποίο θέλουμε να το μειώσουμε από τις 7 στις 5 ημέρες. Ε, προφανώς ε, έχετε πρόβλημα να μετρήσετε ως το 3. Αν ξεφορτωθείτε αυτό λοιπόν σε μία αγορά, θα πρέπει να μετρήσετε καλύτερα, θα πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρο. Είναι μεγάλο λάθος ε, διότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε την οδηγία για το καποτάζ ήταν λάθος το ότι δεν υπόθηκε τίποτα για το τι θα γίνει μετά τη χρήση του καποτάζ. Το φορτηγό θα πρέπει να επιστρέφει στη χώρα του. Αν αυτή η πρόταση υπήρχε αρχή εξ αρχή στο κείμενο, τότε δεν θα ήμασταν εδώ για να διορθώσουμε αυτό το λάθο ε, το οποίο έχει μετεξελιχθεί σε αυτό το τέρας. Δεν έχω ελπίδες ε, για το ότι η οδηγία θα λύσει το πρόβλημα. Ποιος θα διασφαλίσει ότι λειτουργεί οι ε, φορολογικές αρχές, η αστυνομία, κανείς δεν το ξέρει. Είναι ένα ζήτημα οργάνωσης ε, το οποίο θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να κατασκευαστεί. Χρειαζόμαστε λύσεις εδώ και τώρα. Η οδηγία αυτή λοιπόν θα πρέπει να την πάρουμε και να τη σκίσουμε πολύ απλά είναι αδύνατο. Η αστυνομία δεν μπορεί να το ελέγξει. Έχουμε το κείμενο το οποίο λέει ότι οι μεταφορές θα πρέπει λαμβάνουν, να λαμβάνει χώρα ε, στο πιο ορθό μέρος, πιο, ποιος ορίζει τι είναι το ορθό μέρος. Απλά ανοίγουμε την πόρτα σε ε, κακομεταχείριση. Ε, και όσον αφορά την οδηγία καμποτάζ θα πρέπει να διορθωθεί και δεν χρειάζεται αυτή η επιπλέον οδηγία. Ε, βλέπω ότι η οδηγία του καμποτάζ έχει καταστρέψει την αγορά, έχει ανοίξει την πόρτα σε νέες προτάσεις όμως αυτή η μεταφορά για πέντε ημέρες αυτό που, το οποίο καταφέρατε εκεί πέρα είναι να χειροτερεύσετε τις συνθήκες ε, για ε, τις ε, μεταφορές μεγάλων αποστάσεων ε, και έχετε τις ίδιες ανησυχίες ε, για ε, τοπικές μεταφορές όπως και μεταφορές μεγάλων αποστάσεων διότι το φορτηγό μπορεί να περάσει τα σύνορα πολλές φορές ε, και να διανύμει σε διάφορες πόλεις για πέντε μέρες διότι δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των μεταβιβάσεων. Υπάρχουν πολλοί τρόποι λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα στην νομοθεσία. Θα δείτε τις συνέπειες όλου αυτού και η ε, ξεκούραση όσον αφορά την ξεκούραση, ε, είναι όνειρο να λέμε ότι οι ε, οδηγοί θα πάνε σε ξενοδοχείο και θα κοιμηθεί διότι ο οδηγό νιώθει υπεύθυνο για το φορτηγό του, δεν θέλει να το εγκαταλείψει και πόσα ξενοδοχεία έχετε δει εσεί τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν οδηγού με φορτηγά 4 τόνων. Δημιουργείται ένα τέρα λοιπόν. 40 τόνους. Ε, οπότε δημιουργείται ένα τέρας. Σας ε, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιορίσουμε τις παρεμβάσεις μας γιατί το δεύτερο τμήμα των συζητήσεων θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Να παραμείνετε στα τρία λεπτά. Βάντεκαμπ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο λεπτά. Τρία. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι εισηγητής για το θέμα χρόνου οδήγησης και ανάπαυσης ε, και καλό είναι να, να ανταλλάξουμε κάποιες πρώτες σκέψεις. Έχω 7 σχεδόν σημεία αυτή τη στιγμή. Το πρώτο είναι η σχέση μεταξύ των διαφόρων θεμάτων αν εμείς ως ε, Κομισιόν, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο δεν ε, φυλάξουμε την συνοχή μπορούμε να οδηγηθούμε σε καταστροφή. Καλό είναι λοιπόν να παραμείνουν οι ισχυώδεις συγητές και οι συγητές σε επαφή. Στο δικό μου το θέμα η θέση στάθμευσης είναι μεγάλη πρόκληση. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε την ανάπαυση στην καμπίνα του τράκτορα τα Σαββατοκυριακά εάν δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης. Γι' αυτό είναι ακριβώς ασθενής η πρόταση Κομισιόν μας λέει τι πρέπει να γίνει αλλά πώς θα γίνει αυτό και πότε δεν μας λέει τίποτα. Μετά για την αντίδραση. Πρέπει να προσέξουμε λίγο στην αντίδραση ε, και στο ότι βάζουμε συνεχώς τη λέξη κοινωνικό παντού. Η καλή δουλειά και ο μισθός είναι επίσης κάτω κοινωνικό. Κολλάμε παντού την ετικέτα κοινωνικός, κοινωνικός, κάτι το οποίο δεν βοηθάει την απασχόληση στον τομέα των μεταφορών. Μετά το θέμα των ταχογράφων. Εδώ πέρα συμφωνώ με τον πρόεδρο. αν μιλάμε για το 2034 γινόμαστε γελοί. θα πρέπει να δούμε ακριβώς το πώς θα γίνει ο εξυγχρονισμός των ταχογράφων μαζί με την χρηματοδότηση και είχαμε πει πως για τα μεγάλα εμπορικά οχήματα μπορεί να μπει απλά ο ταχογράφος και δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ανταγωνισμού. Με τον Πεντελούντουρεν συμφωνώ για το θέμα του Καμποτάζ και σκεφτόμαστε ούτως ή άλλω στην ομάδα του ΕΛΚ να υπάρξει μια περίοδος cooling down μετά τις ε, πέντε ημέρες απεριόριστου Καμποτάζ. Και τέλος θεωρώ ότι το θέμα ακριβώς του χειρισμού, το τι γίνεται δηλαδή με τον τωρινό κανονισμό ε, και την εφαρμογή του πρέπει να λάβει μεγαλύτερη πρόσοχη στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Θα τελειώσουμε τους συγητές. Η επόμενη ομιλήτρια έχει το λόγο. Παρακαλώ, τρία λεπτά. Η κυρία Μοντέιρο έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή γιατί ήρθε εδώ και μας εξέθεσε το πακέτο κινητικότητας που είναι περίπου περίπλοκο με πολλές θετικές πλευρές, αλλά επειδή είναι πολυσχηδές, από τη δική μας πλευρά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και αυτή είναι μια συζήτηση κομβική σημασίας. Μιλάμε για την εσωτερική αγορά και φυσικά θα πρέπει να δούμε και κοινωνικές ε, πτυχές, αλλά και τα οδικά τέλη. Αυτές οι προτάσεις θα επιτρέψουν τη διασάφιση αμφισημιών καθώς και τα μονομερή μέτρα από ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία θίγουν την εσωτερική αγορά και την διαστρεβλώνουν. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν και να ελεγχθούν από τις αρμόδιες αρχές. Αυτό θα θέλαμε να προτείνουμε γι' αυτό το πακέτο κινητικότητας. Απλά μέτρα, ίση μεταχείριση και σωστή εφαρμογή. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ανισότητες ή ασυμμετρίες, ιδιαίτερα για τις μικρομεσες που αποτελούν την πλειοψηφία των ε, μεταφορέων εμπορευμάτων. Χρειαζόμαστε λοιπόν έμπρακτα εφαρμόσιμα μέτρα. Επειδή είμαι εισηγήτρια σε αυτό το ε, χαρτοφυλάκιο ιδιαίτερα για τα ενοικιαζόμενα οχήματα, θα ήθελα να μιλήσουμε για την χρήση του οχήματος σε άλλο κράτος μέλος για μια ελάχιστη περίοδο τεσσάρων ε, μηνών. Ε, έχει γίνει μελέτη αντικτύπου για αυτή την τετράμινη χρήση. Επίσης, ως προς τους ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές για αυτό το τετράμινο, ξέρουμε ότι οι ελεγκτικές αρχές δρούν διαφορετικά ανάλογα με το κράτος μέλος. Άρα έχουμε ένα θέμα εφαρμογής. Ως προς τα μητρώα των ενοικιαζόμενων οχημάτων, θα ισχύσουν 28 κανόνες που έχει θέσει, είχε θέσει αρχικά η Κομισιόν. Επίσης για την ε, αύξηση άνοδο της ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση της Ρουμανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζονται πολλές διασαφηνίσεις. Ευχαριστώ η κυρία Λουκασέσκα για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πιστεύω λοιπόν το θέμα είναι ότι δεν θα πρέπει να βιαστούμε ε, πολύ με αυτό, διότι είναι δύσκολο να εργαστούμε με αυτόν τον ρυθμό, όμως ε, θα πρέπει να εξαλείψουμε κάθε πιθανότητα ε, κακομεταχείρισης και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να εισάγουμε ε, μέτρα που να βοηθούν τις επιχειρήσεις και εν τέλει θέλουμε οι καταναλωτές και οι ψηφοφόροι μας να είναι ικανοποιημένοι με όλο αυτό. Έχω όμως κάποια ερωτήματα, θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων υπόθηκε αρχικά ότι είναι lex specialis όσον αφορά τις μεταφορές και στη συνέχεια ακούμε ότι το ζήτημα της απασχόλησης θα το διαχειρίζονται άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την απασχόληση. Ε, το, παραδι, το παραδίδει όλο το κομμάτι οι, ε, οι μεταφορές ή ε, ε, η Επιτροπή Απασχόλησης ε, θα ασχοληθεί με το κομμάτι του κομπαντάζ καθώς διαβάσαμε την, την έκθεση αντιτύπου 15 κράτη-μέλη θα είναι ικανοποιημένα ενώ άλλα 13 από την κεντρική Ευρώπη για αυτά οι συνέπειες θα ήταν αρνητικές και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το Καμποτάς αντιστοιχεί στο 2% των μεταφορών οπότε η ιδέα ήταν να αποφύγουμε ε, άδεια ε, φορτηγά και να αποφύγουμε τις ε, περιβαλλοντικές συνέπειες. Τι λοιπόν είναι σημαντικό για την Κομισιόν ενδιαφέρεστε ε, για το περιβάλλον και τα άδεια φορτηγά ή θέλετε να ικανοποιήσετε τα κράτη-μέλη και άλλα να τα εξοργήσετε. Και τώρα όσον αφορά το dumping αυτό είναι μια λέξη ε, που βρίσκουμε στα λεξικά αφορά την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών ε, κάτω του κόστους όμως ακόμα δεν έχω συναντήσει καμία εταιρεία μεταφορών ή οποιαδήποτε επιχείρηση που θα προσέφερε αυτές τις υπηρεσίες κάτω του κόστους, οπότε μιλάμε για ανταγωνιστικότητα. Κατανοώ ότι μερικοί από εσάς αρνείστε να συμφωνήσετε και να το αποδεχθείτε, όμως θα πρέπει να το αποδεχθείτε και αυτό είναι το σύνθημά μου. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα ανάπτυξης μεταξύ των κρατών μελών και διαφορετικά, ε, διαφορετικές τιμές και διαφορετικά κόστη. Ε, καταλαβαίνω λοιπόν την ιδέα, οπότε μην, ε, ε, μην χρησιμοποιείτε έτσι τον όρο αυτόν. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που τηρήσατε το χρόνο σας. Επειδή δεν μπορεί να γίνει πλήρως ή ε, να ολοκληρωθεί η δεύτερη συζήτηση, θα σταματήσουμε με τους εισηγητές και τους σκιώδεις, γιατί θα έχουμε πολύ λίγο χρόνο για τη δεύτερη πτυχή του, της συζήτησης. Έχουμε την κυρία Ντελμόντε τον κύριο Βαμίτελμπουργκ και, την κυρία, και η κυρία Ντέλη και μετά θα περάσουμε στη δεύτερη συζήτηση και η Επιτροπή θα πρέπει να μας απαντήσει. Η κυρία Ντελμόντε έχει το λόγο. Ε, το θέμα είναι ότι θα πρέπει να μιλήσουν οι συγητές και η δεύτερη συζήτηση έχει την ίδια βαρύτητα με την πρώτη. Κύριε Αντελμόντε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχήν συμφωνώ με τον κύριο Βαντεκάμπ γιατί θα πρέπει να φτάσουμε σε συμφωνίες. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στο τέλος της θητείας χωρίς την έγκριση αυτού του πακέτου. Μία πρωταρχική παρατήρηση για τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης που αφορά τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις ανάγκες των τουριστών που πολλές φορές θέλουν να, να σταματάνε σε τακτά χρονικά διαστήματα, να γίνονται δηλαδή στάσεις, συχνότερες στάσεις. Αυτό σε σχέση, σε αντιδιαστολή μάλλον με τα εμπορεύματα. Τώρα, ως Προς τον κανονισμό 561 γίνεται λόγος για έδρα. Εδώ χρειάζονται διευκρινήσεις, γιατί σύμφωνα με το δικό μας δίκαιο υπάρχει διαφορά μεταξύ επαγγελματικής έδρας και ε, έδρας παραμονής. Γιατί εδώ υπάρχει μία διαφοροποίηση. Θα πρέπει λοιπόν να μην υπάρχουν αμφισημίες το 8α σε σχέση με την ανάπαυση, ανάπαυση εκτός φορτηγών, δεν ξέρω κατά πόσο η Επιτροπή δεν έχει διενεργήσει μια μελέτη σε σχέση με υποδομές υποδοχής, γιατί έτσι θα δούμε ποιο είναι και το εμπλεκόμενο ε, κόστος για αυτά τα σημεία ανάπαυσης κοντά στον αυτοκινητόδρομο. Αντί δηλαδή να ε, γίνονται, αντί ε, να ε, γίνεται ανάπαυση μέσα ή κοντά στα φορτίγα. Ως προς το θέμα του καμποτάς θα πρέπει να δούμε τις διασυνοριακές μεταφορές, γιατί το ρυθμιστικό μας πλαίσιο μέχρι τώρα είναι συγκεκριμένο και υπάρχει χάσμα αλλά μπορεί να υπεκφύγουμε και των ρυθμίσεων αυτών. Ως προς τον ταχογράφο, νομίζω ότι θα πρέπει να ε, εφαρμόσουμε τάχιστα αυτό το μέτρο. Τέλος, ως προς τους ελέγχους, ήδη σήμερα γνωρίζουμε ότι πολλές φορές υπάρχουν ε, παραβάσεις χωρίς να υπάρχουν ε, κυρώσει. Ο κύριος Ντέλη έχει το λόγο. Για δύο λεπτά. Uh, Ως ε, νομοθέτες λοιπόν πιστεύω ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα σε αυτό το πλαίσιο και, σε αυτό το πλαίσιο, και όχι απλά να δημιουργήσουμε ε, νομοθεσία έτσι απλά. Το ε, σημαντικό λοιπόν είναι να αντιμετωπίσουμε ε, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες ε, για όλους τους παράγοντες σε όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες και να υπάρξει απλοποίηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταξύ άλλων και επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε ούτως ώστε να έχουμε κανόνες που μπορούν πράγματι να εφαρμοστούν ως σκιώδης ε, του EPPE ε, για το Lex Specialis ε, σχετικά με το πακέτο θα πρέπει να δηλώσω ότι αμφισβητώ την πρόταση της Κομισιόν σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων και επίσης ε, η ε, Επιτροπή ε, η Επιτροπή Απασχόλησης όπως υπόθηκε που ασχολείται με το ζήτημα της απόσπασης ανέφερε τις μεταφορές σε Στην αιτιολογική σκέψη 10. Ε, η ευκαιρία λοιπόν είναι ε, ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την απόσπαση εργαζομένων ε, μέσα στο πλαίσιο της οδηγίας απόσπασης. Υπάρχουν λοιπόν αρκετά ερωτήματα και αμφιβολίες σχετικά με το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ε, το συγκεκριμένο θέμα. Ολοκληρώστε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βαν θα είμαι σύντομος γιατί όλοι έχουν δικαίωμα λόγου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πακέτο κινητικότητας και χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Νομίζω ότι πρόκειται για σωστή ισορροπία μεταξύ αναγκών της αγοράς και προστασίας των οδηγών. Και όταν μιλάμε για τους οδηγούς και χρόνο εργασίας και ανάπαυσης, θα πρέπει να ορίσουμε τα άρθρα 8α και 8β, γιατί γιατί χρειαζόμαστε έναν ευφύ ορισμό και συμφωνώ με τον κύριο Τέλιτσκα ότι πρόκειται για ασφαλή σημεία πάρκινγκ γιατί πολλοί ε, στην ουσία πλήττονται από αυτό, δηλαδή ότι παρκάρουν ε, τα φορτηγά σε όμορες περιοχές ως προς το καμποτάζ οι πέντε ημέρες ε, είναι πολύ. Το τρίμερο θα ήταν ένας καλός συμβιβασμός γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το περιβάλλον. Δεν μπορούμε να έχουμε άδεια φορτηγά που να περιφέρονται στα οδικά δίκτυα και νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την απελευθέρωση της αγοράς. Εδώ μιλάμε και για θέσεις που βρίσκονται σε κίνδυνο, όχι στη Γαλλία και στην Ολλανδία, αλλά στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους Ευρωπαίους πολίτες σε αυτά τα κράτη-μέλη. Άρα ε, μην ακολουθείτε την πολιτική του Διέρη και Βασίλευε. Επίσης, δεν νομίζω ότι μπορεί να εφαρμοστεί στις διεθνείς μεταφορές η οδηγία για τους αποσπασμένους. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, για μένα προσωπικά. Και μιλάμε και για την εφαρμογή και τη θέση και σε εφαρμογή. Όπως είπε ο κύριος Βαντεκάμπ, χρειαζόμαστε ψηφιοποιημένες ε, προσεγγίσεις και ευφύς ταχογράφους. Τώρα, και δεν χρειαζόμαστε ευφυείς ταχογράφους για ελαφρά οχήματα, γιατί αυτό αποτελεί άχθος ιδιαίτερα για την ε, μεταφορά και παράδοση δεμάτων. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κράμερ. Πρώτα απ' όλα θα πω ότι δεν συμφωνώ να αλλάξουμε τους ε, κανόνες ε, στη μέση της συζήτησης. Πρώτα μιλάνε η μεν ε, τρία λεπτά, μετά οι άλλοι δύο λεπτά. Ε, όχι, δεν μπορεί να μιλάμε όλοι λίγο, αλλά όχι η μεν έτσι και οι άλλοι αλλιώ. Λοιπόν, ανταγωνισμός, ναι, ωραία, αλλά να είναι δίκαιος. Δηλαδή, η τιμή της ε, παραγωγής ε, δεν ενδιαφέρει μόνο την επιχείρηση, αλλά και το κράτος. Αν ο επιχειρηματίας δεν πληρώνει το βασικό μισθό, δεν πληρώνει φόρου, τότε πρόκειται για αθέμητο ανταγωνισμό και δεν είναι δυνατόν ο τίμιος να είναι το κορόιδο εδώ πέρα. Ένας νόμος βεβαίως ο οποίος δεν επιβάλλεται δεν έχει κανένα νόημα. Όχι το 2030 επίσης να το εφαρμόσουμε. Η συζήτηση για τους τοχογράφους υπάρχει από το 2013. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα τεχνικά. Είναι ψηλό το κόστος αλλά δεν πάει άλλο με την ε, απάτη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν αν μπει μάλλον με συγχωρείτε το διόδιο θα μετατοπιστούν τα φορτία σε μικρά φορτηγά και σε δευτερεύοντες δρόμους. Επίσης, ο Πέτερ Λούγκρεν έχει δίκιο. Έλεγχη. Δεν επιτρέπεται π.χ. να κυκλοφορούν το Σαββατοκύριακο τα φορτηγά στην Γερμανία. Ωραία, ξεκουράζονται δύο μέρε και μετά πέντε μέρε οδήγηση και μετά ξανά το ίδιο. Και μπορεί να το κάνουν επάπειρον. Επίση, για το βασικό μισθό. Ο Ρουμάνο οδηγό μου είχε πει 8 μήνε οδηγούσα σε Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και ήμουν συνεχώ με στα αυτοκίνητα και μου δίναν 233 ευρώ το ρουμανικό βασικό μισθό. Μιλάμε για σύγχρονη σαβιά, δεν πρέπει να την επιτρέψουμε. Και πρέπει να αλλάξει αυτό συζητούσα χτες ε, με το Γερμανικό Σύνδεσμο Μεταφορέων. Ταχογράφη. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα και να υπάρχουν έλεγχοι. Δεν είναι δυνατόν ο Τίμιος να είναι το χορόιδο, αλλά λένε ναι. Λένε παραδείγματο χάρη είναι μια γερμανική εταιρεία, πάει ανοίγει μια θηγατρική στη Ρουμανία και πληρώνει ρουμανικούς μισθού, ε, πληρώνει 2.000 ευρώ. Και έξοδα επίση, δεν του πληρώνει με, τα έξοδα τα λοιπά, αλλά τα ε, υπόλοιπα τα, το εξοδολόγιο που τους δίνουν δεν είναι φορολογήσιμα. Και εκεί πέρα υπάρχει φορολογική απάτη. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν διαφάνεια, αλλιώ υπάρχει κοινωνικό ντάμπινγκ και δεν το θέλω. Σας ευχαριστώ, κυρία Τάρπαντετ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και εγώ νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι να εκφράσουν την άποψή τους για αυτό το θέμα που είναι ύψης της σημασίας. Αυτό το πακέτο κινητικότητας ήταν απόλυτα αναγκαίο και βρίσκεται ενώπιον μας για να έχουμε μία δίκαιη και ολοκληρωμένη αγορά μεταφορών. Φοβούμε όμως ότι φτάνουμε σε ένα νέο κατακαιρματισμό της αγοράς εργασίας. Η Επίτροπος μας έλεγε ότι υπάρχουν δύο μπλοκ στο Συμβούλιο με αποκλίνουσες απόψεις. Το ίδιο θα γίνει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να λάβουμε μέτρα που να ευεργετούν ορισμένα κράτη-μέλη και να ζημιώνουν άλλα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ναι, έχουμε καθήκον να λάβουμε μέτρα υπέρ των εργαζομένων, υπέρ των πολιτών, αλλά δεν μπορούμε να λάβουμε μέτρα τα οποία θα βγάλουν από την αγορά εταιρείες που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Διαφορετικά θα δημιουργήσουμε ανεργία στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο κύριος Κράμερ μίλησε για την κατάσταση ενός Ρουμάνου που για οκτώ μήνες δούλεψε στην Ευρώπη χωρίς ανάπαυση ουσίας. Αν όμως δου... θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο δούλευε για ρουμανική εταιρεία ή για εταιρεία της Δυτικής Ευρώπης που κάνει τις ίδιες καταχρήσεις. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να επιλύσουμε μέσω νομοθεσίας. Από εδώ θα πρέπει να ξεκινήσουν οι συζητήσεις. Ως προς το δεύτερο μέρος της συζήτησης, επειδή είμαι σκιώδης, θα ήθελα να μιλήσω για τα οδικά τέλη των βαρέων οχημάτων και για να μην μιλήσω δύο φορές θα μιλήσω τώρα. Αναγνωρίζω, αν δεν συμφωνείτε θα επανέλθω αργότερα επί του θέματος, επί του θέματος ε, της φορολόγησης Νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ και δεν ολοκλήρωσα στην Επιτροπή μας. Έχουμε και του συναδέλφους από την Επιτροπή Απασχόλησε. Η κυρία Λαμποβά έχει το Δλαμπάιοβα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ζήτησα τον λόγο στο τέλος για την σκιώδη ε, συγγήτρια στην οδηγία περί απόσπασης εργαζομένων και με όρισαν και η συγγήτρια για το κοινωνικό κομμάτι του πακέτου της κινητικότητας, οπότε θα τα λέμε συχνά στο μέλλον. Με απασχολούν αυτά τα ζητήματα από την αρχή πριν παρουσιάσει την σχετική οδηγία η Κομισιόν πριν από 1,5 χρόνο. Οπότε ε, μπορώ να μιλάω με τι ώρε για αυτά. πάντων, δεν θέλω να το κάνω τώρα. Αν θέλετε λεπτομέρειε, μπορείτε να με ρωτήσετε. Πρώτα απ' όλα νομίζω όπω ήδη αναφέρθηκε από κάποιου συναδέλφου. χρειαζόμαστε την απολύτω σωστή ισορροπία μεταξύ τη ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών και τη προστασία εργαζομένων. Αυτό το οποίο έχουμε τώρα ως πρόταση στην Επιτροπή Απασχόλησης και αναλαμβάνω την ευθύνη ως ε, μία εκ των σκιωδών αφορά περισσότερο την προστασία των εργαζομένων παρά την ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών. Ε, λυπούμε, αλλά ε, είναι ένας συνδυασμός ε, των μελών της Επιτροπής Απασχόλησης, των σκιωδών ενσύτων και οι δε μεταφορές αναφέρονται μόνο στα εκτιμώντας. Πάλευα από την πρώτη στιγμή, βλέπετε εδώ τα αποτελέσματα, πάλευα ή μεταφορές να αναφερθούν στα άρθρα, αλλά δυστυχώς οι σκιώδεις ηγητές δεν το επέτρεψαν, οπότε είναι μόνο στα εκτιμώντας και ανησυχώ ιδιαίτερα για το τι θα γίνει μεταξύ της εφαρμογής οδηγίας περί απόσπασης και της ε, πλήρους εφαρμογής ε, του πακέτου κινητικότητας, γιατί δεν θα είναι ξεκάθαρη η κατάσταση, θα είναι δύσκολη για τις εταιρείε να καταλάβουν τι ισχύει. Δευτέρα λοιπόν, ε, εάν μπορείτε να μιλήσετε με τους ε, σκιώδεις ηγητές της ομάδας σας, ε, θεωρώ εγώ ακόμα ότι η ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών είναι η πιο σημαντική αρχή και δεν με ικανοποιεί ο τελικός συμβασμός. να πω ένα τελευταίο πράγμα. Ε, μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες γιατί γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες της οδηγίας απόσπασης εργαζομένων ανησυχώ ιδιαίτερα για την επικοινωνία. Το ακούτε και εδώ μέσα. Και σας διαβεβαιώ ότι στην Επιτροπή Απασχόλησης είναι χειρότερα τα πράγματα. Είμαστε διχασμένοι, είναι ένα θέμα διχαστικό, υπάρχουν προκαταλήψεις ε, και χρησιμοποιούμε και διατυπώσεις που δεν θα έπρεπε και δεν μπορούμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία στην επικοινωνία. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί κάποιοι λένε ότι γίνεται κατάχρηση από την Τσεχία και τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν ένας Φλαμανδός που είχε στήσει μια τσεχική εταιρεία. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Και έχετε ευθύνη ως Επιτροπή Μεταφορών, γιατί κάπως σας μετέθεσε την ευθύνη η Επιτροπή Απασχόλησης. Ε, και τέλος, αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι πείτε μου τι θέλετε να γίνει με τους φορτηγατζίδες και θα σας πω τι Ευρώπη θέλετε. Η κυρία Βέρνερ θα μπορούσε να μας δώσει ορισμένες διευκρινήσεις αν και όπως σας είπα συνάδελφοι θα πρέπει να εμβαθύνουμε το θέμα αλλά ε, επειδή δεν, θα γίνει, δεν έγινε η ψηφοφορία της έκθεσης του κυρίου Αϊκχάουτ, θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, θα μπορούσαμε να παραμείνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Κυρία Βέρνερ. Thank you very much. It's um, a bit Ευχαριστώ πολύ. Είναι δύσκολο να απαντηθούν όλα αυτά μέσα σε ένα-δύο λεπτά. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσω λέγοντας ότι η Κομισιόν ε, μοιράζεται τις απόψεις που υπόθηκαν από αρκετά ε, μέλη εδώ πέρα και θα πρέπει λοιπόν να ε, δούμε ε, την πρόταση αυτή στο σύνολό της, να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ του περιβάλλοντος, της οικονομίας, της εφαρμογής και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας για να υπάρξει αυτή η ισορροπία και να δημιουργήσουμε κανόνες οι οποίοι θα μπορούν να εφαρμοστούν και να μην τους παρακάμπτει κανείς. Ε, θα ήθελα να ε, ξεκαθαρίσω όσον αφορά την απόσπαση εργαζομένων η οδηγία αυτή ε, η παλαιά του 1996 ναι εφαρμόζεται αυτό το οποίο ε, προτείνουμε εδώ πέρα είναι ένα ειδικό νόμος αποκλειστικά και μόνο για, την, ε, για τις μεταφορές για να για να εφαρμόσει κριτήρια ε, σχετικά με τη μισθοδοσία από την τρίτη ημέρα διεθνών μεταφορών αλλά να εφαρμόζεται άμεσα για λειτουργίες καποτάς. Ε, κάνουμε μια διαφοροποίηση αυτών των δύο και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό το οποίο θα πρέπει να διαφοροποιείται μεταξύ των δύο ε, αυτών ασχέτως του ποιος θεωρείται εσείς είναι ο σωστός αριθμός. Τώρα όσον αφορά την εφαρμογή και το πώς μπορεί να συμβεί αυτό ε, κάτι το οποίο υπόθηκε από την Πρόεδρο. Υπάρχουν αρκετά ε, στοιχεία. Ε, ναι, θα πρέπει να εφαρμόζεται ο ταχόγραφος και όσο, πιο, όσο πιο γρήγορα μεταβούμε στον έξυπνο ταχόγραφο, τόσο το καλύτερο. Κάνουμε μια έρευνα η οποία θα είναι διαθέσιμη το Φεβρουάριο του 2018 και θεωρώ ότι αυτό θα είναι μια σημαντική συνεισφορά και στη συζήτηση σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε σε τεχνολογικό επίπεδο για να εφαρμοστεί πιο εύκολα. Ε, προτείνουμε επίσης ε, περισσότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών, ε, απλοποιούμε τους κανόνες, προτείνουμε ένα μίνιμουμ συχνότητας ελέγχων και ε, δεν ε, ε, ασχολούμαστε με τις κυρώσεις που θεωρούμε ότι ανήκουν στην δικαιοδοσία των κρατών μελών και επίσης η, η απώλεια της καλής φήμης και της άδειας λειτουργίας είναι η βασικότερη, η σημαντικότερη κύρωση για μια εταιρεία. Τώρα όσον αφορά τις συνθήκες ανάπαυσης. Ε, μέσω των απλοποιημένων κανονισμών καμποτάζ ε, δεν θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένο αριθμό ε, δράσεων διότι αυτό είναι δύσκολο να εφαρμοστεί όμως θέλουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών κατά τη διάρκεια των οποίων ε, θα συνεχίζουμε, να εφαρμόζονται οι κανόνες οδήγησης και ανάπαυσης και θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα σημαντικό συστατικό για να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς είναι επαρκές συνθήκες ε, ανάπαυσης σε εβδομαδιαίο επίπεδο. Ε, σε αυτό το πλαίσιο συζητήσαμε και με τα ασφαλή πάρκινγκ για φορτηγά. Θα γίνει μια έρευνα που θα μας επιτρέψει να χαρτογραφήσουμε την κατάσταση ε, και να έχουμε ε, πάρκινγκ τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι οδηγοί ε, και επίσης θα υπάρξει χρηματοδότηση πάνω σε αυτό. Πολλοί από εσάς αναφερθήκατε στην έννοια home θα πρέπει να οριστεί συγκεκριμένα αυτό. βέβαια, από νομικής άποψης δεν είναι τόσο εύκολο. Υπάρχει ένα στοιχείο επιλογής για τον οδηγό, ο οποίος ορίζει ποιο είναι το home, το σπίτι αυτό που θεωρεί σπίτι ε, δεδομένου του γεγονότος ότι δεν έχω χρόνο θα σταματήσω εδώ όμως ξέρω ότι υπάρχουν και άλλα ε, ερωτήματα ε, θα επιστρέψουμε σε αυτά τα ερωτήματα λοιπόν ε, ε, μόλις υπάρξει πρόθεση τώρα όσον αφορά ε, την ενοικίαση αυτοκινήτων οι τέσσερις μήνες συνδέονται με την εποχιακή απασχόληση, εποχική απασχόληση Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να συζητήσουμε γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στη δεύτερη συζήτηση που αφορά τα οδικά τέλη. Ε, Η κυρία Βέρνερ έχει το λόγο και πάλι. προς τις ε, οδικές μεταφορές ε, κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς τα εμπορεύματα και τους επιβάτες και υπάρχουν περιβαλλοντικές ανησυχίες. Θα πρέπει να ασχοληθούμε ε, με το θέμα της μόλυσης του αέρα από τις οδικές μεταφορές και τις μεταφορές γενικότερα σε σχέση με τους στόχους των κλιματικών αλλαγών. Γι' αυτό θα πρέπει να ληφθούν μέτρα τα οποία να είναι σωστά μέσα στα πλαίσια της ε, δίκαιης τιμολόγησης. Ο πληρώνει. Αυτή είναι η απαράβατη θέση μας. Γι' αυτό προτείναμε δύο νομοθετικά κείμενα την οδηγία για την Ευρωβινιέτα για να έχουμε περισσότερη συνοχή στα οδικά τέλη και τον ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό, το ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό ε, σύστημα διοδίων έτσι ώστε να είναι λιγότερο δαπανηρό και για τους χρήστες και για τα κράτη-μέλη. Άρα οι βασικές αλλαγές ως προς την Ευρωβινιέτα έχουν ως εξής. Θα θα ε, διευρύνουμε μάλλον την εμβέλεια για να καλύπτει όλα τα οχήματα. Όχι δηλαδή τα μεγάλα φορτηγά, αλλά και τα μικρά ε, φορτηγά, λεωφορεία και πούλμαν και τους ιδιωτικούς φορείς που συνεισφέρουν στη συμφορήσεις, στη μόλυνση και αφορά όλους τους χρήστες θέλουμε να απομακρυνθούμε με το καταποκοπή ποσό, δηλαδή την κλασική βινιέτα και θέλουμε να έχουμε μία μεταβατική περίοδο και να βασιστούμε στην καταβολή τελών ανάλογα με τη διάνυση απόστασης. Θέλουμε μία απλούστερη εφαρμογή του εξωτερικού κόστους έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει και την ηχορύπανση και την ρύπανση του αέρα. Θέλουμε λοιπόν να αντικατοπτρίζει την πραγματική, τις πραγματικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και για τα ιδιωτικά και για τα εμπορικά οχήματα και να υπάρχει και αποτίμηση του κόστου συμφόρησης και να υπάρχουν τέλη και για την οδική συμφόρηση. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει μία οριοθέτηση για να βρούμε και τις σωστές οδικές ε, λύσεις. Το earmarking θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξο, αλλά θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές σε σχέση με τα αποδεκτά πλαίσια. Ως προς τα ηλεκτρονικά διόδια αντιμετωπίζουμε δύο βασικά προβλήματα. Καταρχήν ε, δεν υπάρχει διασυνοριακή διαλειτουργικότητα που γνωρίζουμε και στο τομέα των σιδηροδρόμων, αλλά αυτός είναι ε, αυτό είναι ένα μεγάλο βάρος. Ήδη το 2013 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να δράσει. Το κάνουμε λοιπόν και ένα άλλο θέμα είναι ότι δεν έχουμε το μέσο για να επιβάλλουμε τα διόδια από παραβάτες, ξένους παραβάτες, αλλοδαπούς παραβάτες και μιλάμε για 300 ε, εκατομμύρια ετησίως. Αυτό θα πρέπει να το δούμε με νομοθετικές ε, πράξεις, δηλαδή την οδηγία διαλειτουργικότητας, όπου μιλάμε για υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών από τους παραβάτες που δεν κατέβαλαν τα διόδια και το δεύτερο μέσο είναι η αναθεώρηση της απόφασης που ορίζει τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά διόδια όπου θέλουμε να άρουμε τα προσκόμματα της εσωτερικής αγοράς. Έτσι θα μπορέσουν οι χρήστες να μεταφέρονται ελεύθερα στην Ευρώπη με, ένα, με μία σύμβαση και μία τιμολόγηση. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει συνάφεια έτσι ώστε να μην περιμένουμε την έγκριση οδηγίας πριν αλλάξουμε την απόφαση. Έχουμε τη σωστή πορεία αλλαγής, Και ξέρετε ότι υπάρχει μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τα διόδια για την άρση των διοδίων στη Γερμανία έτσι ώστε να μην υπάρχει κατακαιρματισμός της αγοράς και μην ξεχνάμε ότι σε αυτό το τομέα μιλάμε για μια βιομηχανία όπου οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατέχουν ηγετικό ρόλο και θεωρώ ότι εάν διατηρήσουμε το πλαίσιο διοδίων τότε θα κρατήσουμε την ε, ηγετική μας θέση. Θα είμαι αμήλικτη ως προς το χρόνο γιατί ξέρετε ότι έχουμε και μία ακρόαση που προβλέπετε. Τρία λεπτά στους δύο εισηγητές και μετά οι ισχυώδεις θα έχουν δύο λεπτά, εντάξει. Δίνω το λόγο καταρχήν στην κυρία Ρεβονταλόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω για την αναθεώρηση της οδηγίας για την Ευρωβινιέτα που θα πρέπει να ανταποκριθεί στην έλλειψη στρέβλωψης των, του ανταγωνισμού μεταξύ των διατροπικών μεταφορών, άρση διακρίσεων μεταξύ χρηστών οδικών αρτηριών, επίτευξη των στόχων της Λευκής Βίβλου έτσι ώστε ο Ριπένον να πληρώνει. Δυστυχώς μόνο το 25% της επικράτειας καλύπτεται από την καταβολή διοδίων. Ε, επίσης, σωστή και καθαρή κινητικότητα, καταπολέμηση της επιδίνωσης των οδικών δικτύων και επίσης σύστημα τελών για τη συντήρηση των οδικών υποδομών. Νομίζω ότι θα πρέπει να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής για όλα τα βαρέα οχήματα, άρση για τα ελαφρά οχήματα και επίσης ορισμός τελών για την υψηλή κίνηση και συμφόρηση και φορολόγηση για τις πραγματικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Έτσι, οι οδηγοί θα πρέπει να κινηθούν προς πιο καθαρά οχήματα και θα πρέπει να δούμε το εξωτερικό κόστος. Η πρόταση της Επιτροπής αφήνει περιθώρια ερμηνείας και γι' αυτό θα προτείνω μέτρα για την ε, εσωτερήκευση του κόστος Δυστυχώς ε, μόνο δύο χώρες έχουν ορίσει αυτά τα τέλη. Ως προς τη μείωση των εσόδων, εάν βασιστούμε στα τέλη αναπόσταση, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα έσοδα χρησιμοποιούνται για την ε, ε ανακαίνιση των υποδομών και επίσης ε, δεν μπορούμε να λαμβάνουμε υπόψη για το όριο του 30%. Επίσης αυτά τα τέλη θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε πιο καθαρές μεταφορές και αυτό αφορά τα διόδια. Τώρα, ερωτήματα προς την Κομισιόν. Πώς αναλύει τον αντίκτυπο των διοδίων σε σχέση με δευτερεύοντα οδικά δίκτυα που δεν διέπονται από τα τέλη αυτά. Έχει επίσης γίνει ανάλυση αντικτύπου για τα διόδια στην περιφέρεια. Πώς θα ληφθούν υπόψη πώς το κείμενο της Επιτροπής θα επιτρέψει στις αρμόδιες αρχές πέρα από τα κράτη-μέλη δηλαδή τις περιφερειακές αρχές, να ορίσουν τέλη υποδομών και τέλος. Γιατί η Επιτροπή θεωρεί ότι τα έσοδα για το εξωτερικό κόστος πρέπει να ενταχθούν στις υποδομές. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τέλη για εξωτερικό κόστος έτσι ώστε οι αρμόδιες αρχές να έχουν μεγαλύτερο εύρος δράσης. Ο κύριος Σαλίνη για τρία λεπτά. σε σχέση με το, τα ηλεκτρονικά διόδια υπάρχουν δύο νομοθετικά πλαίσια. Καταρχήν η οδηγία του 2004 όπου προτίθηκε, προτάθηκε μια αλλαγή με την απόφαση της Επιτροπής του 2009 και το Κοινοβούλιο αναθεωρεί. Ως προς το περιεχόμενο, και όπως είπε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, υπάρχει διεξοδικό πλαίσιο, όμως από το 2004 δεν επικαιροποιήσαμε την οδηγία. Δηλαδή, δεν φτάσαμε σε μία ε, υπηρεσία που να εξασφαλίζει την ε, διαλειτουργικότητα δυστυχώς μιλάμε για ένα εσωτερικό εμπλεκόμενο κόστος που αφορά τα οχήματα και διαφορετικός τρόπος υπολογισμού των διοδίων στα κράτη-μέλη. Ε, η οδηγία προβλέπει να επιληθεί αυτό το ζήτημα. Και από ό,τι φαίνεται οι τεχνολογίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εγγράφονται στην οδηγία. Ενώ στις αποφάσεις λαμβάνουμε υπόψη τις προδιαγραφές που θα ληφθούν υπόψη για την εγγύηση αυτής της δραστηριότητας. Με την αναθεώρηση, δηλαδή επικαιροποίηση της οδηγίας, θα μπορούσαμε καταρχήν να έχουμε μια πραγματική διαλειτουργικότητα και δεύτερον το ακαθόδες ζήτημα των διοδίων, η επίλυσή του. Γιατί ε, δυστυχώς ε, διασυνοριακά δεν καταβάλλονται παντού τα τέλη. Όμως ποιο είναι το πρόβλημα και χρειάζεται φυσικά μία ισορροπία μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Κατά την αναθεώρηση της οδηγίας, ο κατάλογος τεχνολογιών βγήκε από την οδηγία και μπήκε σε ένα παράρτημα, το οποίο θα μπορούσε να τροποποιηθεί από την Κομισιόν με μια κατεξουσιοδότηση πράξη. Άρα αυτό που μας απασχολεί εμάς είναι ότι το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να αποκλειστεί από αυτή τη διαδικασία, γιατί ο κατάλογος της χρήσης των τεχνολογιών είναι ένα απόσπαστο μέρος της συζήτησης. Δεν είναι βοηθητικό, δεν είναι κάτι το επικουρικό. Και αυτό αφορά και το νομικό πλαίσιο που θα μας καλύψει και ως προς τα άλλα συμφωνώ με την Κομισιόν ως προς τα θέματα εργασίας. Ο κύριος Ρικέ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Θα ήθελα να πω ότι λυπάμαι διότι η ελευθερία των μεν καταστέλει την ελευθερία των δε γιατί η προηγούμενη συζήτηση πήρε πολύ χρόνο Όλοι συμφωνούμε ως προς τον απότερο στόχο αυτής της ε, νομοθετικής πρότασης και θα πρέπει οι χρήστες να χρησιμοποιούν αυτά τα δίκτυα αδιακρίτως. Δεν υπάρχει ατέλεια ούτε για τα δίκτυα ούτε για το περιβάλλον. Επίσης, οι χρηματοδοτήσεις θα πρέπει να πάνε στις μεταφορές, γιατί είναι το κέρας της αμάλφιας για το δημόσιο τομέα και ό,τι βγάζουμε ας πούμε από τα καύσιμα πρέπει να πάει στο γενικό προϋπολογισμό. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για την απόδοση των ε, εσόδων γιατί δεν θα πρέπει να γίνουν διακρίσεις και η Ευρωβινιέτα μας δείχνει το εξής. Αν περάσετε μία χώρα ε, ε, μία φορά το χρόνο, καταβάλλετε το κόστος της Ευρωβινιέτας και ας περάσετε από τη συγκεκριμένη χώρα μόνο μία φορά το χρόνο. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξουν αντισταθμίσεις, όπως είπε και η κυρία Ρεβονταλόν. σε σχέση με το αρχικό κείμενο της Κομισιόν. Το earmarking, δηλαδή η επανασύνδεση με τις ε, διατροπικές μεταφορές θα πρέπει να είναι σωστές και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να αποσύρουμε τα ελαφρά οχήματα διότι αφορούν τα δύο τρίτα της κίνησης, της συμφόρησης και της συγχωρήπανσης. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι εκχωρήσεις που, που γίνονται και που δίδονται σε σχέση με την Ευρωβινιέτα. Υπάρχει συνοχή στην πρόταση της Επιτροπής και συνοχή και σε μας. Η κυρία Σενανόβα. Σας eh, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σκιώδης ε, εισηγήτρια για το θέμα αυτό, τα ηλεκτρονικά διόδια και την διαλειτουργικότητα. Χαιρετίζουμε την πρόταση αυτή, έχει την δυνατότητα να επιταχύνει την εισαγωγή διαλειτουργικών συστημάτων διοδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε ακριβώς να παραμεριστούν τα εμπόδια και να βελτιωθεί η ίσπραξη. των διοδίων. Στηρίζω λοιπόν τον εισηγητή στην απόψη του για την πράξη κατεξιοδότηση και για την αλλαγή της ε, λίστας ε, τεχνολογιών στο παράδειγμα. Η δικιά μου ερώτηση είναι να ξέρουμε ποιες τεχνολογίες είναι ξεπερασμένες, ποιες όχι, ποια πρέπει να εισαχθεί κτλ. Το επόμενο μου ερώτημα αφορά της ε, διατάξεις για την εισαγωγή του CITS ε, στα 5,9 GHz. Έχετε κάποια ιδέα για το πώς ε, θα συνδυαστούν αυτές τις τεχνολογίες. Και οπωσδήποτε θα το δούμε αυτό και στο πλαίσιο της συζήτησης για τις προθεσμίες μεταφοράς. Δεν ξέρω αν αρκούν αυτές οι μεταβατικές περίοδοι και αν θα μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε. Για δύο λεπτά ο κύριος Κράμερ. Ναι, ευχαριστώ. Έκανε πολλά πράγματα εδώ σωστά η Κομισιόν, η αρχή ορυπαίνων πληρώνει, οι αποστάσεις, το να υπάρχουν βινιέτες ε, είναι και αντικοινωνικό το να πληρώνει κανείς με 2.000 χιλιόμετρα όσο ένας που κάνει 200.000 χιλιόμετρα και βεβαίως απαιτείται για όλα τα οχήματα. Αν το συγκρίνουμε όμως με τον σιδηρόδρομο, το έχουμε ήδη, είναι ήδη η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ότι πρέπει να πληρωθούν τέλη ε, και βλέπουμε ότι τέλη στους δρόμους πληρώνονται μόνο στο 1% του οδικού δικτύου. Είναι ε, αθέμητος ανταγωνισμός. Τουλάχιστον η Κομισιόν ε, έχει το θάρρος να πει ότι πρέπει να το κάνουμε. Ή Εάν δεν το κάνετε, καταργήστε τα διόδια στον σιδηρόδρομους για να έχουμε μια πολιτική κλίματη, φιλική προς το κλίμα. Αρκεί να το πείτε, το δεύτερο. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ε, έχουν έκπτωση 65%. Κάνουμε το ίδιο και για τα ηλεκτρικά τρένα. Όχι, πληρώνουν όλοι το ίδιο υπάρχει διάκριση στις τιμές μόνο λόγω θορύβου, όχι λόγω καυσίμου. Και εδώ πέρα υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Γιατί μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα και όχι ηλεκτρικά τρένα. Έχουμε ε, μια κατάσταση όπου έχουμε 150 ε, χιλιόμετρα ηλεκτρική γραμμή και μετά 500 χιλιόμετρα ε, κινητήρα στο τρένα. εφαρμογές δεν τις ε, έχετε. Ξέρετε ότι ακριβώς στις περιοχές των Άλπαιων υπάρχουν λόγω των εκπομπών ε, φοβερά πράγματα, λιώνουν οι παγετώνες κτλ. Γιατί δεν το αλλάξατε αυτό παρά το ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και τέλος το earmarking. Ότι θα πρέπει, ε, θα πρέπει να πάνε στο ίδιο μεταφορικό μέσο. Όλοι μιλάνε για shift to rail, αλλά όταν μιλάμε για λεφτά και το πώς θα γίνει, τα έσοδα θα πρέπει να πηγαίνουν ε, στους σιδηρόδρομους. Το κάνουν οι Ελβετοί. Έχουν τριπλάσια διόδια και έτσι φτιάξαν τα τούνελ, ε, τα σιδηροδρομικά. Αυτό πρέπει να κάνετε. Αυτό είναι το σωστό. Ευχαριστούμε κύριε Κράμερ. Κύριε Μπάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω για την Ευρωβινιέτα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για αυτή την παρουσίαση. Συμφωνώ με την ε, κυρία Ρεβονταλόν που μίλησε για το διακύβευμα, το όλο διακύβευμα και τις ε, προκλήσεις. Και η πρώτη της Επιτροπής κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Συμφωνώ με την αρχή ότι ο χρήστης πληρώνει Άρα κάθε χρήστης θα πρέπει να αποδίδει αυτό το κόστος χωρίς καμία εξαίρεση. Όμως η Επιτροπή <coughs> μας δίνει ένα μέσον έτσι ώστε η χρήση των υποδομών να τύχει απόδοσης ε, ενός συγκεκριμένου ποσού για αυτό το σκοπό earmarking. Αυτό το είπε και ο κύριος ε, Κράμερ. Θα προτιμούσα να κινηθούμε προς το ελβετικό πρότυπο. Η Επιτροπή μιλά και για τέλη συμφόρησης. Αυτό είναι ρεαλιστικό, αλλά θα ήθελα το Κοινοβούλιο είναι πιο φιλόδοξο. Έχει νόημα να μιλάμε για κοινέ προδιαγραφές. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να ορίσουν καλύτερα τις ανάγκες τους και τα τέλη αυτά ε, δεν θα πλήξουν τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια μελέτη αντικτύπου. Ως προς τη διαλειτουργικότητα, συμφωνώ με τον συνάδελφο Σαλίνη και με την κυρία Σενάλοβα, θα πρέπει να συνεργαστούμε και θεωρώ ότι η πρόταση της Επιτροπής ε, θα ε, είναι πιο δαπανηρή για τους ε, χρήστες και δεν είμαστε σίγουροι ότι θα γίνουν εκ νέου επενδύσεις προς τις ε, υποδομές. Η κυρία Ταρπαντέλη, για δύο λεπτά ευχαριστώ και ευχαριστώ και την Επιτροπή και για τις δύο προτάσεις θα ασχοληθώ με την πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας και την εφαρμογή οδικών τελών ως προς τα βαρέα οχήματα. Κατανοώ και κατανοούμε όλοι την καταβολή τελών με βάση την απόσταση έτσι ώστε να έχουμε βιώσιμες ε, μεταφορές και φιλικές προς το περιβάλλον. Όμως, έμπρακτα, η πρόσφατη της Επιτροπής ε, Μείωσης των Τελών θα, οδηγεί, θα οδηγούσε σε ανισορροπίες ως προς τους ε, τοπικούς ε, προϋπολογισμούς, γιατί παρεβαίνει στο έργο των Υπουργείων Οικονομικών τι προβλέπει η Επιτροπή για τη μείωση αυτών των ανισοτήτων, ιδιαίτερα για τις χώρες που αυτή τη στιγμή εξαρτώνται από τις οδικές μεταφορές. Με άλλα λόγια, πώς μπορούμε να βρούμε μία μείωση ε, τελών και εισαγωγή τελών ανάλογα με την απόσταση. Ευχαριστούμε την κυρία Ταρπαντέλ, τηρήσατε και το χρόνο σας. Ο κύριος Βαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μια μεγάλη κοινή αποστολή να μειώσουμε το διοξίδιο του άνθρακα, τους ρήπους και να σεβαστούμε την Συμφωνία των Παρισίων. Πρόκειται λοιπόν για την μείωση των ρήπων και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Και χαίρομαι για το ότι η Επιτροπή μας με μεγάλη πλειοψηφία ενέκρινε την έκθεση αυτή για λιγότερες εκπομπές μεταφορές για έναν καθαρότερο κόσμο, για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για τις επόμενες γενιές. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε τις εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα, να είμαστε φιλόδοξοι και το ίδιο ισχύει βέβαια και για την αεροπορία και την ε, ναυτιλία και τι οδικές μεταφορέ. Χαίρομαι Με το ότι σήμερα το πρωί απευθύναμε έκκληση και στην Κομισιόν για να δει το τι μπορούμε να κάνουμε για να σταματήσει η απαλλαγή του ΦΠΑ στα αεροπορικά ειστήρια να δούμε το πώς θα έχουμε ε, τιμιότερη φορολογία, δηλαδή ειδικό φόρο κατανάλωσης στην κυροζήνη και ως κοινωνικά φιλελεύθερος είμαι σίγουρος ότι μπορούν να βοηθήσουν οι ε, μηχανισμοί της αγοράς, δηλαδή η αύξηση των τιμών. Πρέπει λοιπόν να πληρώνει ο καταναλωτής, ο ρηπαίνων, να προστατεύσουμε το περιβάλλον και μέσω έξυπνης καινοτομίας να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Έχουμε έξυπνες και καθαρές μεταφορές, αλλά βεβαίως θα δούμε το τι θα γίνει στην πράξη. Και αν δούμε το γερμανικό σχέδιο περιδιοδίων, είναι περίεργο να πηγαίνει η Κομισιόν προς μια κατεύθυνση μαζί με τη Γερμανία που πηγαίνει ε, μακριά από την πρόταση την αρχική της Κομισιόν. Εκεί πέρα δεν μιλάμε πια για μια πρόταση που είναι ορυπέν πλήρων. Λοιπόν, θα... ωραία αυτά τα οποία βεβαίως λέμε για την διαλειτουργήτα των μηχανημάτων διοδίων, διοδίων κατά το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό γιατί δεν είναι δυνατόν να έχουμε ε, συστήματα τα οποία δεν λειτουργούν τη στιγμή που είχαμε την Ευρωβινιέτα. Πρέπει λοιπόν με την βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι οδικές μεταφορές να περάσουν στον 21ο αιώνα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κράμερ, έχετε μία ερώτηση 10 δευτερόλεπτα. Σύντομα, γιατί μου είπαν ότι η Αυστρία θα μηνύσει την Γερμανία για τα τέλη ε, κατά τον τα τέλη για τα αλλοδαπά φορτηγά. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό, ε, γιατί το δεχτήκατε. Τι θα κάνετε, θα δώσετε τις αρμοδιότητες της ε, Κομισιόν στο δικαστήριο, θα επιμείνετε, τι θα κάνετε ακριβώς. Σας ευχαριστώ, 22 δευτερόλεπτα κάνατε, δεν ήταν άσχημο. Λοιπόν. Η κυρία Βέρνερ έχει στη διάθεσή της 7 λεπτά. plus 4 minutes de tout à περισσότερο από τα τέσσερα που είχατε πριν. Um, uh, Ευχαριστώ πολύ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερος και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερος τον συζητητή αλλά και τους λοιπούς ομιλητές για τη θετική τους αντίδραση ε, πάνω στην ε, πρόταση ε, και επευκαιρίας θα ήθελα από τον συνάδελφό μου Ζουλιά να με βοηθήσει στις δύσκολες ερωτήσεις που μου θέσατε. με τη σειρά που μου ε, τέθησαν, η κυρία Ρεβό ρώτησε τι θα μπορούσαμε ε, να κάνουμε ε, με το δευτερεύον οδικό δίκτυο. Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας θέματα επικουρικότητας. Δεν θα πρέπει να επισέλθουμε πολύ σε αυτό και ε, βέβαια θέλουμε να αποφύγουμε την παράκαψη κυκλοφορίας και ε, να ε, χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία όπου θα υπάρχει δορυφορική παρακολούθηση των διοδίων. Επίσης με ρωτήσατε για τις περιφερειακές περιοχές και αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα σχετικά με την αρχή του ορυπαίνων πληρώνει ε, όσον αφορά τον κύριο ε, Μπαχ ε, θα ήθελα να πω ότι φυσικά και πρέπει να εξετάσουμε το συνολικό άχθος, τα διόδια και την φορολογία που προβλέπεται για τους χρήστες, τους ειδικούς χρήστες. Ακόμα και η χρέωση των διοδίων είναι μια απόφαση των εθνικών κυβερνήσεων ε, μόνο εάν χρεώσουν τότε θα πρέπει να τηρούν την ε, πρόταση ή την ευρωβινιέτα την οποία ήδη υπάρχει. Και φυσικά υπάρχει και το ζήτημα της ε, φορολόγησης που θα επέτρεπε να προσαρμόσουμε το φορολογικό άχθος ή να έχουμε και κοινωνικά ζητήματα τα οποία θα λάβουμε υπόψη μας. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο καλύπτεται ε, από την πρότασή μας. Ε, ένα άλλο σημαντικό σχόλιο που κάνατε είναι ε, σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιούνται τα χρήματα τα οποία συλλέγονται. Είμαστε ανοιχτοί προς συζήτηση ε, θα θέλαμε βέβαια αυτά τα χρήματα να πηγαίνουν προς ε, μέσα βιώσιμης κινητικότητας. Ο κύριος Κράμερ ε, πρότεινε να επεκτείνουμε το γεωγραφικό πλαίσιο για να καλύπτουμε και περισσότερες περιοχές και τα χρήματα μπορούν να μεταφερθούν, να χρησιμοποιούνται στους δρόμους αλλά δεν είναι αναγκαίο. Σε αυτή τη συζήτηση λοιπόν σχετικά με το πώς αντιμετωπίζονται άλλα είδη Μεταφορών η Κομισιόν ε, κάνει μια έρευνα ε, σχετικά ε, με τα εξωτερικά κόστη όλων των τρόπων μεταφορών οπότε δεν έχει ολοκληρωθεί όμως οπότε δεν μπορώ να λάβω θέση πάνω σε αυτό θα είναι μια, πρόταση, μια συζήτηση την οποία θα κάνουμε στο μέλλον ρωτήθηκαν επίσης ζητήματα μετάβασης ιδιαιτέρως ε, με τις ε, παραχωρήσεις και τα συστήματα ε, βινιέτας και θα πρέπει να βρεθεί μια λύση πάνω σε αυτό και να λάβουμε και το χρονοδιάγραμμα υπόψη μας. Τέλος, αλλά όχι έσκατο, σχετικά με την τεχνολογία η οποία προτείνεται να προσαρμοστεί με πράξη κατεξουσιοδότηση το ε, θέμα εδώ δεν είναι να περιορίσουμε τις τεχνολογικές πλευρές. Ε, καταλαβαίνω ότι αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι για τη λειτουργία του συστήματος. Όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι συγκεκριμένες προσαρμογές θα πρέπει να γίνονται γρήγορα. Ε, διότι γνωρίζουμε πώς ε, πηγαίνει η νομοθετική διαδικασία κάθε φορά που υπάρχει ένα ε, νέο τεχνολογικό ε, επίτευγμα στην αγορά. Θα θέλατε εσείς να προσθέσετε κάτι. τώρα όσον αφορά τα γερμανικά διόδια, γνωρίζετε ότι η ε, Κομισιόν έκλεισε ε, το ε, ζήτημα και προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε μεταξύ της Γερμανίας και της Αυστρίας σχετικά ε, με το άρθρο 259. Σεβόμαστε την απόφαση της Αυστρίας να μεταφέρει το ζήτημα στο δικαστήριο, όμως θέλουμε να έχουμε μια ευρωπαϊκή λύση, ούτως ώστε τέτοιες διφωνίες να αποτελέσουν παρελθόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Βέρνερ. Δεν έχουμε γενέθλια εδώ. Ευχαριστούμε τους διερμηνείς που παρέμειναν ε, πέντε λεπτά επιπλέον. Θα σας ξαναδώ τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου στις ε, τρεις ε, στη γενή ακρόαση με την Επιτροπή Απασχόλησης για την κοινωνική πτυχή της κινητικότητας και τους άλλους, τους υπόλοιπους θα τους δω στις 9 9 Νοεμβρίου. Α, ως προς την ψηφοφορία θα σας στείλω mail γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ούτε αίθουσα ούτε ώρα. Αναβλήθηκε η ψηφοφορία εδώ και δύο ώρες. Ε, δεν είμαι μάγος. Καλό απόγευμα. Γεια σας.